Uh, so, ladies Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην ε, πρώτη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας υπό την ε, δικιά μου Προεδρία και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να δουλέψω στη θέση αυτή και ε, είχαμε σήμερα το 2,5 ώρες ε, πολύ σημαντική συνεδρίαση με τους συντονιστές και θα αναφερθώ αργότερα ε, στο θέμα αυτό αφού ακούσουμε τον Επίτροπο και αφού οργανώσουμε την ημερήσια διάταξη. Θέλω όμως να καλωσορίσω τους εκπροσώπους εδώ και ιδίω αυτού οι οποίοι είναι νεοεκλεγέντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τους ευχαριστήσω που επέλεξαν την Επιτροπή μα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πείρα του στην εργασία της επιτροπή μα. Θέλω επίση να ευχαριστήσω και ολουσμένους συναδέλφου που ήρθαν από άλλε επιτροπέ για να προσφέρουν την πείρα του και ιδιαίτερω του αντιπροέδρου μου την κυρία Κόχολα, τον, ε, τους, ε, την κυρία Κόχολα, τον κύριο Βερνιό, την κύριο Κόμη και τον κύριο Γκρέχ. Θα ήθελα όμως ε, καταρχήν να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει η ημερήσια διάταξη η οποία είναι κάπως διαφορετική από αυτήν την οποία είχατε δει και θα ήθελα να ξέρω εάν συμφωνείτε ε, με τις τροποποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Ωραία. Τότε έτσι θα προχωρήσουμε και η τελική μου ο παρατήρηση που είναι σημαντική προτού καλέσω τον κύριο Φερχόιγγεν να μας μιλήσει είναι να τονίσω μία αλλαγή, δηλαδή ότι η συνεδρια μας θα τελειώσει πιο νωρίς, προβλέπουμε να τελειώσουμε στις 5.30 διότι μετά υπάρχει ε, μία δεξίωση που οργανώνεται από τη Σουηδική Προεδρία και θα έρθουν ε, οι εκπρόσωποι του Σουηδικής Κυβερνήσεως που θα μας μιλήσουν αρχίσουν αύριο και σας καλούν όλους να συμμετάσχετε. Θα παρούξω λοιπόν να μην φύγει κανείς σας πιο νωρίς νομίζοντας ότι τέλος ε, η συνεδρίαση αλλά να υποφεληθείτε από αυτή την ευκαιρία. Οπότε κάνω τη δήλωση αυτή στην αρχή της συνεδριάσεως. Εάν λοιπόν τώρα συμφωνείτε, είναι ιδιαίτερη χαρά με εμένα να ε, σας καλωσορίσω να καλωσορίσω και τον κύριο Φερχόιγγεν διότι έχουμε συνεργαστεί ε, στενά όσο ήμουν συντονιστής για το ΕΛΚ και έχει προσφέρει την ε, πείρα του στο στην ε, Επιτροπή μας και στα προγράμματά μας έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα προγράμματα και είναι μεγάλη χαρά για μένα να ε, καλωσορίσω εδώ τον Γκίντερ. Ξέρω ότι θέλει να μας παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο θέμα που είναι η ε, οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών και θα ε, ε, ακούσει μετά οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να απευθύνετε σχετικά με την, ε, τον τομέα των αρμοδιοτήτων του. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα έχουμε μια πολύ ενεργή και ζωντανή συζήτηση και ξέρετε ότι έχει ήδη ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών οπότε φροντίστε να τραβήξετε την προσοχή του γραμματέα και δίνω τώρα το λόγο στον Γκίντερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάκομ. Η πολιτική της χώρας μου ούτως ή άλλως ε, με υποχρέωνε να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα η θέση μου αυτή και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι ευρωβουλευτές, δική μου είναι η χαρά που παρίσταμε εδώ ως φιλοξενούμενό σας σε αυτή την πρώτη τακτική συνεδρίασή σας και θέλω πρώτα να συγχαρώ θερμά τον Μάκομ Χάμπορ για την εκλογή του ως Προέδρου αυτής της Επιτροπής και όλους σας να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στην Ευρωβουλή ως Ευρωβουλευτές. Σας εύχομαι μια επιτυχή κοινοβουλευτική θητεία σε όλους σας παρότι αυτό κάπως θλίβει το ότι ο χρόνος που, από, που κοινού, από κοινού σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα είναι πιθανότατα πολύ περιορισμένος. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο, ποια θα είναι η διάρκεια αυτή, αλλά σας διασφαλίζω ότι θα ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας εγώ και οι συνάδελφοί μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την τελευταία ημέρα. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι την τελευταία ημέρα μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ε, για να δοθεί απάντηση. Ποια θα είναι η τελική τελευταία έκβαση και ποια θα είναι αυτή η διάρκεια δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή αλλά προτούμε κάποια συγκεκριμένα νομοθετικά θέματα δραστηριοτήτων να απασχοληθούμε. Κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για την κατάσταση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Ναι, στην ακμή ακριβώς, στον κολοφόνα αυτής της ε, οικονομικής κρίσης ε, που έχει, μας έχει πλήξει όλους ε, και που ζήσαμε σε μια περίοδο που αρχίζει να τελειώνει ή να απηχεί περισσότερο αυτή η οικονομική κρίση. Τουλάχιστον η εικόνα αυτή είναι μετά τις θερινές διακοπές κάπως πιο αισιόδοξη, κάπως πιο θετική από ό,τι πριν από τις θερινές διακοπές. Είχαμε δραματικές εξελίξεις όπως όλοι γνωρίζετε στον τομέα όσον αφορά για παράδειγμα τα ελεύθερα επαγγέλματα και τις ε, δραστηριότητες σχετικά. Τα σημαντικότερα πλήγματα 2008-2009, πρώτο τρίμηνο 2009, κανένας από αυτούς που γνωρίζω και με μεγάλη πείρα στην πολιτική, στην οικονομία δεν είχαν ζήσει μια τόσο ταχεία συρρήκνωση κατάπτωση, καταποντισμό της ευρωπαϊκής οικονομικής ε, δραστηριότητας και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την κατάρρευση δεν ήταν η έλλειψη ανταγωνιστικότητας ή αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ούτε η ελλειψη της ενίας εσωτερικής αγοράς υπό το οικονομικό ε, πλαίσιο της τάξης των πραγμάτων που είχαμε εμείς δημιουργήσει. Ήταν αντίθετα το αποτέλεσμα μιας ε, θα έλεγα χωρίς έλεγχο εκρηκτικής ανάπτυξης που κατάφερε τελικά να υπεκφύγει εθνικών ελέγχων, δηλαδή όσον αφορά ελέγχους σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες του οικονομικού κόσμου. Και θα ήθελα να πω ότι τώρα που αρχίζει η εικόνα να δείχνει λίγο καλύτερα, δεν θα πρέπει να διστάσουμε ή να φοβηθούμε να συναγάγουμε με σαφήνεια τα συμπεράσματα με κάθετο τρόπο και κατηγορηματικά από αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι προφανώς ο συνδυασμός όλων των μέτρων που λάβαμε συνεισέφερε ε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτή την κρίση από ό,τι υποθέταμε στην αρχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει η ασφάλεια, η βεβαιότητα ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Και βλέπω ότι Πότε παρά σήμερα τα αναγκαία αυτά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και θα πρέπει να είμαστε κάθετοι και με σαφήνεια προ όφελο τη ενιαία εσωτερική αγορά κιόλα και προ όφελο ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό που θέλουμε είναι να αποφύγουμε. Να αποφύγουμε για άλλη μια φορά να οδηγηθούμε σε αυτή την γιγαντιαία διαστάσεων αποστεγανοποίηση ή αποσύνδεση των οικονομικών αγορών από την πραγματική οικονομία. Και δεν βοηθάει καθόλου να έχουμε για μια χρονιά σε μια, να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε 2% του τζίρου παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίμακα να έχουμε ανταπόκριση στην πραγματική οικονομία και 98% μόνο αναφορά σε, ε, εικονική ε, οικονομική πραγματικότητα. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, διότι είδαμε πόσο άμεσες είναι οι επιπτώσεις μιας οικονομικής κρίσης ε, στις, στα οικονομικά, στα δημοσιονομικά, στις τράπεζες, Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που βρίσκονται στο περιθώριο της ε, χρεοκοπίας ή της μη φερεγγιότητας ε, οικονομικά, διότι η οικονομική κρίση έδωσε αφορμή να μην παραταθούν ε, δυνατότητες αποπληρωμής δανείων με τα οποία είχαν επιφορτιστεί και έτσι να υπάρχει και συρρήκνωση κερδών επιχειρήσεις που ήταν σύγχρονες και ήταν αποτελεσματικές και με επιτυχία λειτουργούσαν στις αγορές Προ όφελο ακριβώ αυτών των επιχειρήσεων πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα του οικονομικού τομέα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή έχουμε στην πραγματική οικονομία στην Ευρώπη είναι πράγματι η διασφάλιση πιστώσεων. Και αρκετές φορές έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για τους πιο διαφορετικούς λόγους και η αντιμετώπιση και πρόληψη κινδύνων, η επικέντρωση σε άλλες δραστηριότητες οδήγησαν τελικά η διασφάλιση πιστώσεων και δανείων και από μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πιέζεται, να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση και να υφίσταται πιέσεις καταφέραμε όσο καλά μπορούσαμε να το κάνουμε να έχουμε μια διεύρυνση των δανείων, των πιστώσεων τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες για μια αντιστάθμιση τη κατάσταση. Αλλά οι δυνατότητε επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι περιορισμένε και την πλήρη λειτουργία ενός ε, ενιαίου ε, συνολικού συστήματος τραπεζικού δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει αυτές τις δραστηριότητες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και έτσι έχουμε τώρα αυτή την τεράστια σημασία που βλέπουμε να δίνεται σε αυτή τη δράση. Αν είχα μια επιθυμία, Πρόεδρε, που θα μπορούσε να υλοποιηθεί, θα έλπιζα και θα ευχόμουν οι Ευρωπαίοι να τα καταφέρουν στην σύνοδο της λέσχης των 20 κρατών να είναι πιστικοί και δραστήριοι στα συστάσεις τους και να μιλήσουν με μία φωνή, με μία ενιαία φωνή. Αυτό είναι το πιο αποφασιστικό αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται τώρα νομίζω, περιτεύει να αναφερθώ στην συνολική εικόνα σφαιρικά. Απλά και μόνο σύντομα να σας ενημερώσω και να πω ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις ε, στην παραγωγή τις είδαμε στην παραγωγή μετάλλων και επεξεργασίες μετάλλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανοβιομηχανίας και παραγωγής μηχανών. Ωστόσο σταθεροποιείται τώρα, αντισταθμίζεται αυτή η τάση, αυτή η κατάσταση. Και από μήνα σε μήνα στις συγκρίσεις που κάνουμε βλέπουμε για πρώτη φορά ότι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μια σχετική αύξηση. Αλλά σε σύγκριση ετών από έτος σε έτος βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική συρρήκνωση και θα υπάρξει ακόμα μια σειρά ετών που θα χρειαστεί θα το χρειαστούμε αυτό ως χρονική πρόπτικη ώστε να φτάσουμε στην παραγωγή του 2007 κάποτε στο μέλλον. Και πρέπει αυτό να το επισημάνω. Είναι σημαντικό νομίζω για την κοινοβουλευτική σας επιτροπή, για τις κοινωνικές ε, οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Ποιες θα είναι. Τώρα ήδη με αυτή την, ας το πω έτσι, απόσβεση αυτής της κρίσης θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογές διαρθρωτικές σε διάφορους οικονομικούς τομείς και δραστηριότητες. Τώρα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να λάβουν εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία ώστε να προσαρμοστούν οι διαθρώσεις τους και να υπάρξει προσαρμογή σε ένα επίπεδο παραγωγής και αυτό υποχρεωτικά θα οδηγήσει σε, μια, σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ανέργων που θα δημιουργηθούν λόγω αυτών των προσαρμογών. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και θα πρέπει έγκαιρα τα μέσα να λειτουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε κάποια μέσα, κάποια εργαλεία με τα οποία μπορούμε να αντισταθμίσουμε και να κάνουμε κάτι. Για παράδειγμα, το, η σκόπιμη και αποτελεσματική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαθωτικών Ταμείων, των μέσων που αφορούν τις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την υποστήριξή τους. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ως εύρος μέτρων που μπορούμε να υιοθετήσουμε και να εκτελέσουμε. Όμως συνολικά η κατάσταση η, η κατεύθυνση, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της οικονομίας μας πρέπει να παραμείνει σε ένα σταθερό πλαίσιο. Αυτή η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίζεται από την αναγκαιότητα μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής επανάστασης που πρέπει να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρωθεί με τις επιπτώσεις που θα οδηγήσει σε μια, για παράδειγμα, παραγωγή και αποτελεσματικότητα στην χρήση της ενέργειας, αποτελεσματικότητα αλλά και αηφορία και αηφορία όχι μόνο οικολογικά πράγμα το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οικονομικά είναι επιταγή αυτό να επιτευχθεί, διότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που οι παγκόσμιες αγορές απαιτούν. Και βλέπουμε ότι οι μεγάλες κοινωνίες που είναι ανεπτυγμένες έχουν μια χόρταγη ζήτηση και ανάγκη για αγαθά που επιτρέπουν σε αυτές τις κοινωνίες να συνεχίσουν την αναπτυξιακή τους πολιτική και πρέπει να την συνεχίσουν, να μπορέσουν να την συνεχίσουν διαφορετικά η κοινωνική πίεση θα ήταν αφόρητη. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και το περιβάλλον να διασφαλίζεται και να προστατεύεται. Εδώ ανοίγεται, διανοίγεται για μας ως Ευρωπαίους μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα προτέρημα και είμαστε προπομπή. Είμαστε σαφώς ε, η προπομπή, η πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα παγκόσμια. Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε αν πραγματικά πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό και πολύ δραστήριους ε, ανταγωνιστές, ως συναγωνιστές ε, και για τις νέες αλλαγές και πρωτοβουλίες από πλευρά της Αμερικανικής νομοθεσίας πρέπει να συλλάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Βλέπουμε εδώ το δυναμικό και τις δυνατότητες όσον αφορά τους Αμερικανούς και υπάρχει και η διαφορά κλίμακα. Αν δει λοιπόν κανείς ε, τι γίνεται σε σχέση με χρεοκοπημένες επιχειρήσεις ε, εκεί, κανένας δεν έδινε ούτε μια δεκάρα, ούτε ένα σέντ για το μέλλον των ε, μεγάλων αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Σήμερα, λίγες εβδομάδες μόνο αφού πέρασαν από τη διαδικασία χρεοκοπία λάμπουν πάλι με αυτοπεποίθηση και αστράφτουν και ιδιαίτερα σε σχέση με General Motors. Αναφέρομαι και στη General Motors γιατί διαφορετικά θα επανέλθω στη συνέχεια άμεσα σε αυτό, σε αυτήν, στη συνέχεια. Αυτό δείχνει τις ικανότητες και δυνατότητες των Αμερικανών, τι μπορούν να κάνουν αν θελήσουν να κάνουν κάτι. Και κατά τα άλλα έχουν και αυτή την μακροπρόθεσμη ε, ε, διάσωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας που διασυνδέεται με τη δική τους ε, κατεύθυνση που ακολουθήθηκε. Και αυτή που είχαμε εμείς με το ΚΑΣ 21 του 21ου αιώνα που είχαμε υιοθετήσει, προσαρμογή όλων αυτών με την, τον νέο ανταγωνισμό που πλευρά είπα. Να αναφέρω ακόμα δύο πράγματα αν, αν επιτρέπετε. Το πρώτο, το ερώτημα, η ενιαία εσωτερική αγορά σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Λειτουργήσε ή όχι. Είχαμε σίγουρα, ιδιαίτερα στον τύπο της χώρας που γνωρίζει καλύτερα ο πρόεδρος, στα αγγλοσαξονικά μέσα του τύπου είχαμε έντονες προειδοποιήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση προστατευτικών τάσεων, προστατευτικών τάσεων από πλευράς της Ευρώπης και σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία που αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο στην υπηρετική Ευρώπη υπήρχαν έντονες προειδοποιήσεις. Αν δούμε όμως σήμερα την πραγματικότητα πρέπει να πω λοιπόν τότε ότι πάρα πολύ λίγες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έκαναν καν προσπάθεια με την βοήθεια προστατευτικών μέσων ή μέτρων να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και να διασωθούν υπήρξαν κάποιες ρητορικές εχμές όσον αφορά τον προστατευτισμό. Αυτό δεν το αμφισβητώ, δεν μπορώ να το διαμφισβητήσω. Ήταν πολλές φορές έντονες αυτές οι αιχμές προστατευτισμού. Όμως το σύστημα αποδείχθηκε αρκετά ικανό και δυνατό και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήταν αρκετά δυνατά και ισχυρά ώστε μια αναζωογόνηση του οικονομικού προστατευτισμού να αποφευθεί. Εδώ τώρα θέλω να επανέλθω σύντομα για το θέμα της General Motors. Αυτό το ερώτημα, αυτό το ζήτημα για το μέλλον της, ε, των ευρωπαϊκών θηγατρικών επιχειρήσεων της General Motors θέτει ένα θεμελιώδες ζήτημα για την ενιαία εσωτερική αγορά. Η General Motors έχει ε, θέσεις παραγωγής σε σχεδόν 12, μια ντουζίνα ευρωπαϊκές χώρες. Όμως επικεντρώνεται σε μία επιχείρηση στην Γερμανία ιδιαίτερα. Και βλέπουμε ότι η γερμανική κυβέρνηση καταρχήν προσπάθησε να το αντιμετωπίσει ως δικό της πρόβλημα, καθαρά γερμανικό. Και προσπάθησε λοιπόν να ακολουθήσει μια πολιτική που την έδρα επιχειρήσεων στη Γερμανία θα την διασφάλιζε για την προοπτική υπέρ αυτών των επιχειρήσεων στη Γερμανία. Είπαμε ευθύ εξ αρχή εμεί ότι εμεί δεν πιστεύουμε, δεν θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να βοηθηθεί υιοθετώντα, αποκλείοντα έναν ανταγωνιστή από την αγορά και αν κάποιος ανταγωνιστής έχει μια πιθανότητα να ανταγωνιστεί, πρέπει να του δίνεται αυτή να ανταγωνιστεί. Και τώρα για το πώς η General Motors στην Ευρώπη θα μπορούσε να διατηρηθεί, δεν ήταν το μόνο αυτό ζήτημα. Λέγαμε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, λέγαμε, και όχι καθαρά γερμανικό μόνο. Τα επιμέρους μέτρα που θα υιοθετηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται και να είναι ε, συμβατά και να συνάδουν με τα ευρωπαϊκά μέτρα και σταθμά. Και όλα πρέπει να γίνονται σε απόλυτη διαφάνεια, ώστε όλες οι εμπλεκόμενες χώρες να μπορούν τα συμφέροντά τους να τα διασφαλίζουν με τον πιο διαφανή τρόπο. Μέχρι τη σημερινή ημερομηνία, μέχρι σήμερα, το καταφέραμε αυτό να το πετύχουμε. Για την έκβαση όλης αυτής της υπόθεσης δεν μπορώ να προδικάσω το τι θα γίνει, γιατί οι τελευταίες αποφάσεις δεν είναι θέματα μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης, ε, ευρωπαϊκής κυβέρνησης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ο ιδιοκτήτης που έχει την κυριότητα αυτής της επιχειρήσεως είναι εκείνος που θα, έχει τον τελευταίο λόγο. Και η General Motors και η, το Αμερικανικό θησαυροφυλάκιο, δηλαδή η Αμερικανική οικονομία. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν από τις επαφές, επαφές μαζί μας ότι άσχετα ποια θα είναι η λύση που θα υιοθετηθεί τελικά, οπωσδήποτε θα εμείνουμε και θα επιμείνουμε ότι δημόσια κονδύλια μόνο τότε θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αν και όταν οικονομικά κάτι τέτοιο θα είναι σκόπιμο να γίνει. Δηλαδή, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις που θα εγκριθούν ή εγγυήσει που θα εγκρινόντουσαν, μόνο υπό αυτή την πτυχή θα τις εξετάσουμε. Είναι συμβατά και συνάδουν όλα αυτά ως αποτέλεσμα, με ένα βιώσιμο οικονομικό αποτέλεσμα ως τελικό στόχο. Και αρκετές φορές ε, δημόσια ανέλαβα πρωτοβουλία να επισημάνω δημόσια ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο οι επιδοτήσει ή ενισχύσει απαγορεύονται. Απαγορεύονται χωρί καμιά αμφιβολία. Μόνο κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται τέτοιε δράσει. Δεν είναι ω κανόνα κάτι το οποίο επιτρέπεται, αλλά μόνο ω ε, ε, ε, ως συγκεκριμένη εξαίρεση. Δεν επιτρέπονται λοιπόν ενισχύσεις. Ενισχύσεις για παράδειγμα για την διάσωση μιας επιχείρησης ή για την αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης με πολιτικά αιτήματα. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση αρχές της, ε, του έτους σε, μια, ένα κράτος μέλος ε, όπου πολιτικά αιτήματα είχαν συνδεθεί με, κάτι τέτοιες, με κάποιες τέτοιες ε, επιδοτήσεις ή αιτήματα ενισχύσεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθετα αρνήθηκε. Αυτό ισχύει όμως και για όλους κάθετα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και να διασφαλίζει ότι οι πολιτικέ τέτοιε δεν επιτρέπεται να συνδέονται, να συναρτώνται σε, στην υιοθέτηση τέτοιων μέτρων. Όμως, Εν τέλει, ένας απολογισμός για την λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε αυτή την κρίση είναι θετική έκβαση αυτού του, του απολογισμού. Θα έλεγα ότι η ενιαία εσωτερική αγορά συνεισέφερε από πλευρά τη με τον τρόπο της, ώστε η κατάρρευση συνολικά να μην είναι τόσο έντονη συνολικά όσο είχε προβλεφθεί. Και αυτό είναι νομίζω σημαντικό για τις επιχειρήσεις, διότι ήταν διαφορετικές οι εξελίξεις σε σχέση με τις διαφορετικές μας χώρες και τις επιχειρήσεις ανά χώρα. Είναι καταρχήν ενδιαφέρον να δει και να πει κανείς ότι σε κάποιες χώρες, σε κάποιες χώρες σημειώνεται ανάπτυξη πάλι, οικονομική ανάπτυξη, όπως στην Πολωνία για παράδειγμα. Είναι μια αγορά, η αγορά της Πολωνίας εκεί και σημειώνει ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, για την οικονομική κατάσταση, αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το ερώτημα για τα προγράμματα τα οικονομικά των κρατών μελών και τα μέτρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσθετα υιοθετήθηκαν με τριοπαθέστερης κλίμακας πρέπει να ομολογήσω τι κατάφεραν να ε, αποφέρουν αποτέλεσμα από αυτά τα, να έχουμε ως αποτέλεσμα από αυτά τα μέτρα. Ένα όμως μπορούμε ήδη σήμερα να πούμε προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να έχουν άμεση επίπτωση, γιατί διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα να υιοθετούνται και να εκτελούνται. Πρέπει να έχουν τέτοια μορφή και τύπο εκτέλεσης ε, και τέτοιο χρονικό πλαίσιο, ώστε η άμεση επίπτωση να είναι δεδομένη και πρέπει να έχουν τέτοια μορφή στην ε, εκτέλεσή τους, ώστε να μην παρακολύονται οι αναγκαίες οικονομικές προσαρμογές, να μην διατηρούνται δηλαδή κάποιες δομές και διαθρώσεις που μακροπρόθεσμα δεν θα είναι α, ανταγωνιστικές και πρέπει να παίρνουν τέτοια μορφή αυτά τα προγράμματα ώστε οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές και οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας να μην διακυβεύονται συνολικά, πράγμα το οποίο προανέφερα. Το δεύτερο τώρα, το δεύτερο για αυτή την κρίση, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να είναι σεβαστοί. Και έτσι νομίζω αν λάβουμε όλα αυτά υπόψη τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα αρκετά θετικά. Αν δείτε την οικονομική συγκυρία υπάρχει μια ε, διατήρηση, διασφάλιση στους τομείς εκείνους που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξυγχρονισμός δικτύων, πάσης μορφής, ε, εξυγχρονισμός υποδομών, αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης ενέργειας, απόδοσης ενεργειακής αποδοτικότητας, ε, το άλλο σημείο, πόσο γρήγορα θα έχουν επιπτώσεις αυτά τα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και πόσο αηφόρα θα είναι, δεν μπορώ να το απαντήσω ακόμα σήμερα. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία. Είδα κάποια στοιχεία για τη Γερμανία τα οποία δεν μπορώ να τα πιστέψω ακόμα. Ένα κλάσμα, ένα μικρό κλάσμα των προβλεπόμενων κονδυλίων για αυτά τα προγράμματα που έχει διατεθεί σε αυτή την κατεύθυνση αν πει κανείς ε, από πού θα καλυφθεί αυτή η ανάπτυξη ε, θα ήταν δύσκολο να συναρτηθούν αυτά τα δύο. Λοιπόν, θα έπρεπε να πω ότι δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Έχει όμως τεράστια σημασία να γνωρίζουμε για την ε, ενιαία εσωτερική αγορά πια μακροοικονομικά φορολογικά μέσα από αυτά που έχουμε για την ενιαία εσωτερική αγορά θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικά. Για το, το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης με κριτικό πνεύμα αντιμετωπιζόντουσαν ε, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να απόσχουν από το να παρεμβαίνουν και να ε, επεμβαίνουν με την ε, ορθή θα έλεγα κατεύθυνση των οικονομικών προγραμμάτων θα μπορούσαμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει όμως προσεκτικά να παρατηρήσουμε τις εξελίξεις και ιδιαίτερα συνετά και προσεκτικά να τις αξιολογήσουμε στο μέλλον. Επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια και παρατηρήσεις όσον αφορά την γενική οικονομική κατάσταση και εξέτασή της. Διότι δεν γνωρίζω ακόμα πόσες ευκαιρίες θα έχουμε μια τέτοια, για μια τέτοια συνάντηση και ανάλυση στο μέλλον. Ε, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Από αυτά που τα τελευταία χρόνια ως ε, επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμαθα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών της θητείας μου, θα έλεγα η ενιαία εσωτερική αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ κάτω των δυνατοτήτων της ακόμα. Είναι ένα πολύ καλό θετικό πράγμα η δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη, σε αύξηση της ευημερίας. Εξακολουθούμε να έχουμε υπερβολικά πολλούς φραγμούς και προσκόμματα ε, ψυχολογικής ε, μορφής, πολιτικής, νομικής ε, συγκυρίας που το πλήρες δυναμικό δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί αυτή τη ενιαία εσωτερική αγορά και βρισκόμαστε κάτω από αυτό το δυναμικό είναι σαφώς καλύτερα, καλύτερη κατάσταση για την ενιαία ε, εσωτερική αγορά αγαθών. Εδώ όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν την Ευρώπη ως την δική τους αγορά, την δική τους εγχώρια εντό εισαγωγικών ευρωπαϊκή αγορά. Και όσον αφορά για την ε, ε, αποστολή την ανάπτυξη αυτών των αγαθών σε αυτή την αγορά πολλά προσκόμματα έχουν απαλληφθεί. Υπάρχουν όμως και πάρα, πολλά, ε, πολλές, πάρα δυνατότητες, ένα ιδιαίτερο δυναμικό που θα πρέπει να το παρακολουθήσετε με ιδιαίτερη, να παρακολουθηθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία σε, ε, που έχει υιοθετηθεί για την παροχή υπηρεσιών και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω πολύ σύντομα μόνο να αναφερθώ σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία μας απασχολούν από κοινού. Ο πρόεδρος ήδη είχε προαναγγείλει ότι θα έλεγα κάτι για την οδηγία για την καθυστέρηση πληρωμών στις συναλλαγές. Είχε υποβληθεί πριν από τις θερινές διακοπές αυτή η οδηγία και ως συνεισφορά για την αντιμετώπιση της ε, ε, οικονομικής αρνητικής συγκυρίας. Ένα στοιχείο θέλω να αναφέρω. Αν όλες οι πληρωμές ε, στην Ευρώπη γινόντουσαν έγκαιρα, τότε 86 δις ευρώ θα είχαν επιπλέον ε, ως ε, επιπρόσθετο ποσό στη διάθεσή τους ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι μικρό ποσό. Ήταν εκείνο το οποίο είχε στη διάθεσή της για πέρσι, για παράδειγμα, η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν πρέπει να υποτιμάμε λοιπόν αυτή την, αυτό το μέγεθος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις διασφαλίζεται εναντί άλλων επιχειρήσεων. Εδώ ένας στόχος πληρωμής ως τελική προθεσμία συμφωνείται σε μια τέτοια συναλλαγή μέσα σε αυτό το χρονικό όριο που ο παραγωγός δίνει στον πελάτη για εξόφληση υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλωμένων μερών αυτό, αυτή η προθεσμία ή και νομικά από πλευράς της νομοθεσίας προβλέπεται και επιβάλλεται ο παραγωγός ε, ε, αναμένει μέχρι τέλους αυτής της προθεσμίας το αργότερο να έχει αποπληρωθεί, να έχει εξοφληθεί. Αν γίνει η πληρωμή, αν δεν γίνει μέσα στο πλαίσιο αυτό η πληρωμή, τότε κάνουμε λόγο για καθυστέρηση. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκε ώστε οι καθυστερήσεις πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα. Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία μπορούν για παράδειγμα νομοθετικά κατοχυρωμένοι τόκοι και με βάση ε, ε, συγκεκριμένα επιτόκια να επιβαρύνουν εκείνον που καθυστερεί να πληρώσει. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρότι άρχισε να ισχύει αυτή η οδηγία 35 ΕΟΚ, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, ε, στις συναλλαγές μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και επιπλέον πέρα από αυτά, Υπάρχει, υπάρχουν αποδείξεις, σαφή τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία ότι σε μια ολόκληρη σειρά κρατών μελών οι συμβατικές αυτές οι υποχρεώσεις εξόφλησης ε, σε σχέση με συναλλαγές με το δημόσιο, με κρατικές αρχές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις. Αν σκεφτείτε ότι ένα τρίτο όλων των παραγγελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραγγελίες του δημοσίου ή κρατικών υπηρεσιών, ε, τότε πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα μπροστά μας. Αυτά τα δύο προβλήματα οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις και κολλήματα εμπόδια στην ενιαία αγορά και σε μια φάση συρρήκνωσης ύφεση εντείνεται ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Αυτές οι πρακτικές είναι, ε, υπονομεύουν την φερεγγιότητα και την ρευστότητα των επιχειρήσεων και δυσχεραίνουν τη δημοσιονομική διαχείριση. Οι καθυστερήσεις πληρωμές λοιπόν υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που δεν έχουν και κάποιο μαξιλάρι για απόσβεση τέτοιων προβλημάτων ή κραδασμών ώστε να αντέξουν μια τέτοια περίοδο θα έλεγα ξηρασίας ή ε, τέτοιων προβλημάτων. Οι καθυστερήσεις έχουν ιδιαίτερες δημιουργούν ιδιαίτερες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις μας μια κατά τα άλλα βιώσιμη ανταγωνιστική επιχείρηση μπορεί να υπονομευθεί και να γονατίσει και να καταστραφεί διότι έχουμε μια λυσιδωτή αντίδραση αλυσωτή αντίδραση ξεκινά από την παραγωγή το, την ε, ε, υπονόμευση της εξόφλησης ε, και την αξιοπιστία της και όλα αυτά αυξάνονται μια και η πρόσβαση στα οικονομικά μέσα σε πιστώσεις και δάνεια δυσχεραίνονται μέσα σε μια τέτοια κρίση τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που έχουν σημαντική, ε, μεγάλη σημασία και πρέπει να έχουν ιδιαίτερα διευκολυμένη πρόσβαση σε πιστώσεις και δάνεια ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν από τις δυνατότητες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Έχουμε μια νέα τέτοια διατύπωση της οδηγίας 2035 τώρα που ε, υποβάλλεται από πλευράς μας και που πρέπει να ασφαλίζει, να διασφαλίζει και να αυξάνει την αποτελεσματικότητα ε, των μέτρων αυτών καταπολέμησης ε, των καθυστερήσεων στις εξοφλήσεις, στις πληρωμές και στις συναλλαγές αυτές. Και έτσι λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με το εξωτερικό και εσωτερικό κόστος. Κέντρο βάρους είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο χωρίς να επεμβαίνουμε. Ιδιαίτερα όσον αφορά το ε, δημόσιο τομέα, τον κρατικό τομέα. Να πούμε αυτό κάθετα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για καθυστερήσει σε τέτοιε πληρωμέ από τον κρατικό τομέα ή το δημόσιο. Κανένα, κανένα τέτοιο επιχείρημα, κανένα τέτοιο καμιά τέτοια δικαιολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κανένα δεν μπορεί να πει Α, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατότητα να εξοφλήσουμε αυτέ τι παραγγελίε που είχαμε δώσει. Και όταν λοιπόν το δημόσιο δεν πληρώνει, ε, τότε πρόκειται για μια οικονομική διαχείριση εις βάρος κατά κανόνα μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να προστατευτούν και να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα διότι το δημόσιο, ο τομέας ο κρατικός είναι ο σημαντικότερος πελάτης τους και δεν μπορούν να ε, αμυνθούν εναντί μιας τέτοιας ε, καταστρατήγησης. Θέλουμε λοιπόν το δημόσιο να υποχρεώνεται τέτοιου είδους εξοφλήσεις ή λογαριασμούς που για την παράδοση εμπορευμάτων ε, συνεπάγεται εξόφληση μέσα σε 30 μέρες. 30 ημέρες να εξοφλούνται. 30 ημέρες. Μπορούν και πιο πριν να εξοφλούνται βέβαια, αλλά μετά από αυτές 30 ημέρες έχει δικαίωμα ο ε, πιστωτής να έχει επιπρόσθετο ποσό 5% για τις, ε, την καθυστέρηση που προκαλείται στην εξόφληση αυτή. Γι' αυτό συνειδητά το έχουμε διαμορφώσει με αυτό τον ε, ε, ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο ώστε να είναι αποτρεπτική η επίπτωση, το αποτέλεσμα αυτού του κανόνα ώστε να μην αξίζει πια για κανέναν στο δημόσιο τομέα να καθυστερεί την εξόφληση τέτοιων πληρωμών από το δημόσιο έναντι των επιχειρήσεων. Αυτό ταυτίζεται κατά τα άλλα με μέτρα που μια ολόκληρη σειρά κρατών μελών υιοθέτησαν πολλά κράτη-μέλη είχαν ε, αναγνωρίσει και είχαν δει ότι αν επέλυαν αυτό το πρόβλημα θα συνεισέφεραν με σημαντικό τρόπο για την βελτίωση της κατάστασης και μια ολόκληρη σειρά κρατών μελών λοιπόν. Στο πρόσφατο παρελθόν υιοθέτησαν τέτοια μέτρα ώστε ο δημόσιος τομέας να μπορεί ταχύτερα να εκτελεί αυτές τις πληρωμές. Αυτό ισχύει για την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τις κατοχώρες, την Πορτογαλία και πρόσφατα ε, προλίγου και για την Ιταλία παραμένει ένα εθελοντικό μέσο αυτή η οδηγία, καθότι δεν υποχρεώνει τους συμβαλόμενους ε, να απαιτήσουν τέτοιου είδους επιπρόσθετες, ε, επιπρόσθετους τόκους, αλλά διανοίγει μια τέτοια δυνατότητα. Κατά τα άλλα δεν είναι δυνατόν δεν, σε περίπτωση ε, ε, συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων δεν δημιουργούνται εξαιρέσεις. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μεταξύ ε, υπηρεσιών του δημοσίου να διανοίγονται δυνατότητες. Δεν αξίζει να συζητάμε αν αυτό είναι σωστό ή όχι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν θα θέλαμε κάτι άλλο να κάνουμε θα έπρεπε να πούμε ότι θα επεμβαίναμε στο συμβατικό πλαίσιο διαμόρφωσης των υποχρεώσεων των συμβαλωμένων και δεν θα μπορούσαμε με ένα τέτοιο τρόπο παρεμβατικό να είμαστε αποτελεσματικοί. Γι' αυτό ο το κύριο βάρος αυτών των ε, μέτρων βρίσκεται εκεί επικεντρωμένο και εκεί ε, συναντάται όπου αφορά το δημόσιο τομέα, ο τομέας ε, ο κρατικός και για την ενεργοποίηση τέτοιων απαιτήσεων δημιουργούνται πλαίσια τα οποία διευκολύνουν την απέτηση αυτών των ποσών. Πρέπει όμως να το πούμε αυτό ότι με πολιτικά μέσα ή μέτρα η ηθική δεν μπορεί να βελτιωθεί όσον αφορά τις ε, συναλλαγές. Ιδιαίτερα όταν έχουμε σχέσεις μεταξύ ενός ε, ισχυρότερου και ενός πιο αδύναμου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι στην οικονομική ζωή όταν δημιουργούνται τέτοιες περιπτώσεις πρέπει με το αντίστοιχο πλαίσιο να επιλύονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν όσο ταχύτερα θεωρούμε ότι ε, θα υιοθετηθεί αυτό το μέτρο, τόσο ταχύτερα θα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα από αυτό. Και επιτρέψτε μου εν τέλει να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι θα το χαιρετίζαμε αυτό αν πριν από τα τέλη του 2009 θα είχαμε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να κάνουμε λόγο για έναν απολογισμό αυτού του εγχειρήματος μείωσης αντιμετώπισης ε, της γραφειοκρατίας ιδιαίτερα όσον αφορά το γραφειοκρατικό κόστος το οποίο προκαλείται για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσω της επιπρόσθετης γραφειοκρατίας. Αυτά είναι μέτρα υπέρ της ενιαίας εσωτερικής αγοράς στον τελικό του στόχο. Και εδώ βρισκόμαστε πλήρως ενεργοποιημένοι και προσπαθούμε να προαγάγουμε αυτό το στόχο και η δική μας Επιτροπή θα προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Πάντα με τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή το συζητούσα αυτό το εγχείρημα και θα ήθελα και ευχαρίστω να συνεχιστεί αυτό. Εδώ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα θα ήθελα να αναφέρω που κάποιες ανησυχίες δημιουργεί. Ήδη πέρυσι το Δεκέμβριο είχαμε προτείνει οκτώ ανεδαφικές παροχημένες οδηγίες από τον τομέα του, της ενιαίας εσωτερικής αγοράς να απαλληφθούν οδηγίες που δεν αξίζει τον λόγο να διατηρηθούν και που μπορούν να απαλληφθούν επειδή οι προηγούμενες ρυθμίσεις ε, για αυτούς τους τομείς ε, μέσω διεθνών ε, ρυθμίσεων έχουν ήδη αλλάξει. Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους αντιδράσεις. Είδαμε λοιπόν σε σχέση με την ταχεία απάλληψη αυτών των οδηγιών να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ταχύτερα. Θα ήταν σίγουρα κάτι το ενδιαφέρον να θα μπορούσαμε να ε, ολοκληρώσουμε αυτό το στόχο. Εν τέλει θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω τούτο. Θα ανταποκριθούμε σε εσά και στα αιτήματά σας και με μια πρόταση που την οφείλω σε εσά ε, Σβάμπ. Και έχω πρέπει να πω τύψη συνείδηση, κύριε Σβάμπ ότι δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το εγχείρημα. Όμως τα χρονικά πλαίσια και οι πιέσει δίνουν μια ευκαιρία παρόλα αυτά πρέπει να πω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε, αυτή την, ε, σε αυτό το δικό σας ε, αίτημα. Το, την οδηγία, τη νέα πρόταση για τα, τους γεωργικούς ελκυστήρες, τα τρακτέρ, τον Οκτώβριο θα μπορέσουμε να σας την παρουσιάσουμε. Και είναι αυτό το δυσχερέστατο, για αυτό το δύσκολο θέμα, νομίζω μπορώ να σας καθησυχάσω, βρίσκεται στη δική σας αρμοδιότητα και έτσι θα μπορέσει να διευθετηθεί τον Οκτώβριο. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος διεξοδικότερα μπόρεσα να αναφέρω το, για το πακέτο για την φαρμακοβιομηχανία. Είναι κάτι που είναι αυτονόητο ότι ενδιαφέρει και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή σας και πρόκειται εδώ απλά για το εξής. Για την ενιαία εσωτερική αγορά, για την φαρμακευτική βιομηχανία, την φαρμακοβιομηχανία που έχει μεγάλη σημασία για την ενιαία εσωτερική αγορά να επιτύχουμε ένα υψηλότατο βαθμό ασφάλειας, ασφάλειας για τους πολίτες μας για αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, εδώ επακούμε στα όσα είχα να αναφέρω. Ο κύριος Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι είμαι πρόθυμος να λάβω θέση και να απαντήσω σε όλα τα θέματα που αφορούν το δικό μου χαρτοφυλάκιο και τις δικές μου ε, οι ευθύνες ως τομέα αρμοδιοτήτων. Χαίρομαι λοιπόν για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτές τις ερωτήσεις ανταποκρινόμενος. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την ε, πολύ ευρία ομιλία που παρουσίασε και δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσουμε να ακούσουμε μία πολύ σημαντική και ε, εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των ε, οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε, διαπιστώνουμε ότι η οικονομία της Ευρώπης είναι σε καλή κατάσταση, παρόλο που ορισμένοι δεν συμφωνούν. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών, είμαι βέβαιος ότι θα σημειώσουμε όλοι το ποσό των 86 ε, δισεκατομμύρων δισεκατομμυρίων που θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν εάν όλες οι δημόσιες αρχές κινούνται εντός των προθεσμιών που τους έχουν ταχθεί. Και νομίζω ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο επικοδομητικά. Προς πληροφόρησή σας θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρόκειται να λήξουμε το θέμα αυτό σήμερα, διότι αύριο το απόγευμα θα έχουμε μία συζήτηση και θα έχουμε μία ιδέα της στρατηγικής η οποία προτείνεται. Ελπίζουμε δε ότι η, Ευρωπαϊκή, ότι η Επιτροπή μας θα συμφωνήσει ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε ε, να αξιολογήσουμε την ε, μελέτη των επιπτώσεων προτού προχωρήσουμε στη διατύπωση μέτρων. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε χρόνο τώρα και έτσι έχω 7 ομιλητές μέχρι στιγμής. Δεν έχω ελέγξει. Υπάρχουν ε, άλλοι, ε, όλοι οι συντονιστές θέλουν να παρέμβουν, δύο συντονιστές μέχρι στιγμής ζητούν το λόγο. Εάν λοιπόν θέλουν να μιλήσουν οι συντονιστές, τους παρακαλώ να ξεκινήσουν, αλλά θα ξεκινήσω με τη σειρά που έχουν ζητήσει το λόγο οι διάφοροι ευρωβουλευτές. Υπάρχουν εννέα ενδιαφερόμενοι και θα κάνουμε δύο ομάδες των τεσσάρων για να έχουμε μία συζήτηση εντωμεταξύ. Για τους πρώτους πέντε ομιλητές έχω την κυρία Γκέπχαρτ, την κυρία Σάλντε Μπόζερ, ε, την κυρία Μόζερ, την κυρία Μπάνια και ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στην Εύελιν Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γκούντερ για την πολύ καλή ανάλυση την οποία ακούσαμε και για το πλαίσιο το οποίο μας παρουσιάστηκε για τον οικονομικό χώρο μέσα στον οποίο συζητάμε εδώ γιατί η εσωτερική αγορά της Ευρώπης είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι καλό να ακούμε πιο εμπεριστατωμένα περί τίνος πρόκειται από ό,τι μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Εδώ τίθεται και το ερώτημα τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πολύ σημαντικές. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να προσθέσω μία ιδέα σε αυτά που είπες Γκούντερ, δηλαδή ότι αυτές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας και για μας σοσιαλδημοκράτες είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος γιατί αυτή είναι βασική στόχη τους οποίους έχουμε. Δεν θέλουμε μόνο να πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις αλλά οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν καλά για να ευημερούν και οι πολίτες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Επ' αυτού λοιπόν ε, στα πλαίσια ε, με το σχέδιο αυτό των, ε, της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών δεν έχω ασχοληθεί λεπτομερών αλλά ξέρω ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητες διότι έχουν πολλές εκκρεμότητες δεν έχουν επαρκή ρευστότητα και το, ο αριθμός που ανέφερες και τον οποίο πρώτη φορά άκουσα είναι εξωφρενικός 86 δισεκατομμύρια. Δεν ήξερα ότι μιλάμε για τόσα μεγάλα νούμερα. Είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Και καλό είναι να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είναι επίσης βασικό αυτό το οποίο τόνισες. Δηλαδή ότι ουσιαστικά οι δημόσιες υπηρεσίες φταίνε. Και αυτό είναι πολύ βασικό, διότι πάρα πολλές ε, πληρωμές ε, ε, και πολλές οφειλές ανέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες και εγώ ίδια ξέρω περί την ομιλούμε στο θέμα αυτό γιατί με έχει θίξει. Είναι πολύ βασικό. Το άλλο που είναι πολύ βασικό και που θα ήθελα εδώ να μην αποκρύψω είναι ότι στην ε, προεκλογική περίοδο στη Βάντι Βουτεβέργη ε, πήγα σε πολλές ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες οι οποίες ομόφορα μας είπαν και παραπονέθηκαν ότι δεν πληρώνονται εγκαίρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί υπάρχουν χρέη και κρεμότητες οι οποίες είναι σημαντικές και φαντάζομαι ότι το έχει λάβει υπόψη ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύνεται και αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα, διότι υπάρχουν απλά προγράμματα, ιδίω μικρά, τα οποία είναι στα όρια της χρεοκοπία, διότι δεν τα βγάζουν πέρα πλέον. Σε αυτό το θέμα έχω άλλη μία παρατήρηση. Ότι δηλαδή χρειάζομαι μία πιο σαφή διευκρίνηση. Γιατί εμείς, ε, εάν μπορούμε να υποχρεώσουμε το δημόσιο αλλά όχι τον ιδιωτικό τομέα, διότι νομίζω το σημείο αυτό το πέρασε πολύ ελαφρά. Βεβαίως υπάρχει μία ελευθερία συμβάσεων, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι τόσο ισχυρές όσο οι μεγάλες και αυτές πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα και τα μέσα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς να τιμωρούνται επειδή δεν μπορούν να καταβάλουν χρήματα. Άρα ε, είναι το σημείο στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Η κυρία Σάλντερ Μόζερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μερικές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Για όλα όσα μας είπε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική ανάλυση της κατάστασης ε, και συμφωνώ με πολλά από όσα ε, είπατε. Συμφωνώ όμως ε, και με την Εύελιν. Αν μπορούσαμε να αναφερθούμε καταρχάς στις προδιαγραφές ρευστότητας. Δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περιοριστικοί στους κανόνες μας αυτή τη στιγμή. Είναι καλό για να υπάρχει χρηματοδότηση, να υπάρχουν δάνεια από τις τράπεζες ώστε να υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Αλλά πρέπει να θέσουμε και κάποιους κανόνες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε να περιμένουμε να περάσει λίγο ακόμη περισσότερο η οικονομική κρίση για να μπορέσουμε να θέσουμε πιο αυστηρούς περιορισμούς. Ενδεχομένως ε, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα ε, να έχουν οι επιχειρήσεις μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να ε, καλύψουν τα χρέη τους. Και αναφέρομαι κυρίως στις δημόσιες αρχές και στον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αυτό ήταν ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω. Έχω τώρα και ένα ερώτημα να θέσω. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να εξυγχρονιστεί και να επισπευθεί ε, η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τις δουλειές τους και πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες αλλαγές. Έχω και ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ναυπηγείο στη δική μου περιοχή, το οποίο είπε ότι θα πρέπει να κλείσει γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με ε, την αυπηγική δραστηριότητα στην Ασία. Και θα ήταν χρήσιμο να μπορούμε να πούμε στους πολίτες, στους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους βοηθήσει ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής. Δεν είναι παρκές να πούμε, α ναι, έχουμε διαρθρωτικά κονδύλια. Αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να μπορούμε να τους πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί και ότι κάνει συγκεκριμένες ιδιαίτερες προσπάθειες για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και κάτι ακόμη, και είναι και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, Η ερώτηση που ήθελα να κάνω ακούγοντα όλοι σα την ανάλυση. Κατά την προεκλογική εκστρατεία μου ετέθη εμένα προσωπικά αυτό το ερώτημα. Με ρώτησαν λοιπόν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, υποβάλει την πρόταση αυτή. για τα φάρμακα τα οποία διδόνται κατόπιν ιατρικής συνταγής, κατόπιν συνταγογράφησης. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει υποβληθεί αυτή η πρόταση από πλευρά Επιτροπή. Θα μπορούσα να θέσω και άλλα ερωτήματα, αλλά για την ώρα αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ράπτη τώρα έχει το λόγο, που είναι και νέο μέλος ε, από την ε, Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια κύριε Πρόεδρε. Ε, με το θέμα της οδηγίας, την οποία μας αναπτύξατε, ασχοληθήκαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα σε μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εμπορίου. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και νομίζω ότι έχει σημασία να σας μεταφέρω μια αποστροφή του λόγου του. Ο πρώην Έλληνας Επίτροπος και πρώην Ευρωβουλευτής για δύο θητείες, ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος είπε πάρα πολύ απλά ότι η οδηγία αυτή υπάρχει μεν στα χαρτιά, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Και όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά συμβαίνει και κάτι ακόμη, το οποίο βεβαίως δεν συμβαίνει μόνο στη δική μας χώρα. Αντιμετωπίζεται η κατάσταση της καθυστέρησης των πληρωμών με τις λεγόμενες υπερτιμολογήσεις. Άρα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, αυτό το 5% με το οποίο θα χρεωθεί ο δημόσιος τομέας πώς μπορεί να περπατήσει παράλληλα με τις υπερτιμολογήσεις οι οποίες δεν έχουν σταματήσει. Και α, παίρνοντας αφορμή και από τα όσα υποστήριξε προηγουμένως η συνάδελφος με το θέμα της φαρμακοβιομηχανίας, είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί στην Ελλάδα πάρα πολύ τα νοσοκομεία. Και α, μιλώντας το ίδιο μήκο κύματος ακριβώς με την Εύελιν, το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά αυτή την περίοδο που η ανεργία μας κοιτάζει προς τα πάνω. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ακούσω πώς το αντιμετωπίζετε και παράλληλα θα ήθελα να μου πείτε ε, γιατί αισθάνομαι ότι είστε εξαιρετικά αυστηρός, έτσι όπως μας περιγράψατε την ένταση με την οποία θα πρέπει να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν τα προγράμματα, τα οικονομικά, οι οικονομικές συμβουλές από την πλευρά της Επιτροπής, αλλά δεν είστε το ίδιο πιεστικοί όσον αφορά οδηγίες σαν αυτή που συζητούμε τώρα. Το λέω αυτό και κλείνω, διότι στην Ελλάδα έχουμε έντονο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο πάρα πολύ σύντομα θα μας οδηγήσει σε εκλογές. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Um, um... Ευχαριστώ, κύριε Ράπτη. Ε, ευχαριστούμε πολύ που μας, ε, ε, που μας είπατε όσα μας είπατε και κατόπιν της εμπειρίας που έχετε αποκτήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για όλα όσα μα είπατε ειδικότερα όσον αφορά την ε, καθυστέρηση των ε, πληρωμών και τη σχετική οδηγία. Καταλαβαίνω και συμφωνώ με την πρότασή σας, αλλά δεν ε, μου αρέσει πάρα πολύ το εθελοντικό σύστημα. Προτιμώ το υποχρεωτικό με τις 30 ημέρες και την επιπλέον χρέωση. Ίσως να μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα Εγώ είμαι πολύ υπέρ της ίσης μεταχείρισης, ειδικότερα όσον αφορά την ε, εσωτερική αγορά και θα ήθελα να μου πείτε και εσείς ποια είναι η άποψή σας. Ε, θα ήθελα να μου πείτε επίσης ποια πιστεύετε ότι είναι τα εμπόδια που παραμένουν στην εσωτερική αγορά. Επίσης συνεργαστήκαμε όσον αφορά τις, ε, τους συντελεστές για την επιπλέον χρέωση. Συζητήσαμε πέρσι και με τον κύριο Σφαμπ για ε, κάποιες ηλεκτρονικές ε, συσκευές, ε, όπως για παράδειγμα το σύστημα ESP. Και θα ήθελα να σας υποβάλω και σήμερα ένα σχετικό ερώτημα σε σχέση με αυτό. Σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν διαφορετικά συστήματα συναγερμών και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε από κοινού με το σύστημα ESP, θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να μπορούν να υπάρχει ένα σύστημα υποχρεωτικής, ε, υποχρεωτικού εντοπισμού μέσω του GPS ε, των ε, αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί, γιατί έτσι το 99% των οχημάτων που έχουν κλαπεί μπορούν να βρεθούν εντός κάποιων μηνών. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. πάρα πολύ ασφαλή συστήματα συναγερμού σημαίνουν ότι δεν είναι εύκολη κλοπή των οχημάτων. και έτσι δεν θα υπάρχει και πολύ μεγάλη δυνατότητα carjacking. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της κατασκευής, της ε, συναρμολόγησης του αυτοκινήτου μπορούμε να το λάβουμε αυτό υπόψη γιατί μερικές χιλιάδες ευρώ κοστίζει και ούτως ή άλλως έχουμε δορυφορικά συστήματα, υπάρχει η τεχνολογία, ο συντονισμός είναι μόνο ε, το ζήτημα και ούτε καν αυτό ενδεχομένως η θέληση μόνο να είναι ε, το μόνο που μας λείπει γιατί τότε οι καταναλωτές μπορούν να πούν ότι έχουν πραγματικά μια εσωτερική αγορά και ότι αισθάνονται Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, ε, είναι μια νέα γωνία, μια νέα οπτική γωνία η δική σου, όπως πάντα. Το σύστημα που θα ε, μας βοηθούσε πάρα πολύ είναι να υπάρξει επικύρωση τώρα, να μην περιμένουμε άλλο. Ο Μισελ Μπανιέ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Τεν Φερχόγγεν ότι χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που τον βλέπω και πάλι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, όσον αφορά ε, την οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών σε εμπορικέ ε, συναλλαγέ. Θα ήθελα να του θέσω ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με τα διδάγματα τα οποία εμεί ε, μπορούμε να πάρουμε από την οικονομική κρίση και ποιο είναι ο αντίκτυπο ειδικότερα στι επιχειρήσει. Όσον αφορά την οδηγία, κάνετε μία πρόταση εναρμόνιση των ε, προθεσμιών ε, εμπορικών, πληρωμών των εμπορικών συναλλαγών ε, εντό 30 ημερών. Εντάξει, αλλά υπάρχει μία de facto διαφορά ε, λόγω των διαφορετικών συστημάτων των κρατών μελών ε, και δεν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο προβάδισμα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ε, δημόσιες. Όταν μιλάω για δημόσιους φορείς θα ήθελα να συμφωνήσω με την Ελληνίδα συνάδελφο που ε, αναφέρθηκε σε ένα πολύ συγκεκριμένο ε, θέμα και μίλησε και για διάφορες κοινωνικές δομές, κάτι το οποίο βεβαίως θα δικαιολογούσε Γκίντερ κάποια ε, συστήματα, κάποιες παρεκκλήσεις, κάποιες εξαιρέσεις. Τώρα, όσον αφορά το, αφορά το 5% αποζημίωσης, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετά σημαντικό για να έχει τόσο αποτρεπτικό χαρακτήρα όσο θέλουμε δηλαδή να αποτρέψει ε, να, απο, να αποτρέψει όχι μόνο την δυνατότητα καθυστέρησης των πληρωμών, αλλά γενικότερα τις συναλλαγές. Δεν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Βεβαίως ε, υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα σε πολλές χώρες και σε χώρα που γνωρίζω εγώ όλος ιδιαίτερος. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξουν οι συνθήκε για να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, όχι όμω μόνο για αυτέ. Κάτι ε, το οποίο ε, θα σημαίνει ότι πρέπει τις ε, οικονομίες μας, να τις κατευθύνουμε ε, στις, ε, στους τομείς που αποτελούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό όχι λόγω της ενισχυμένης συνεργασίας που την έχουμε μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας, γιατί αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει να βρεθεί ένας τρόπος κινητοποίησης των οικονομιών μας στο πλαίσιο των διδαγμάτων που θα πάρουμε από την κρίση. Ε, να υπάρχει ε, διαφάνεια, να υπάρχει έλεγχος, ε, ενδεχομένως να μπορούμε εκ των προτέρων να κάνουμε κάποια πράγματα, η κινητοποίηση κάποιων αποταμιεύσεων στις, στους στρατηγικούς τομείς του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, λοιπόν, θα σε αφήσω να ασχοληθεί με αυτές τις ε, ερωτήσεις και ε, μετά θα προχωρήσουμε στην ομάδα από τον κύριο Σβάπ, την κυρία Στήλερ και άλλους δύο ομιλητές. Θα κλείσω την, ε, τον κατάλογο των ομιλητών όταν θα έχει ομιλήσει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ε, παρακολούθησα τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Εύελιν, η Εύελιν όντως έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων για την Ευρώπη και εμένα με εξέπληξε ο αριθμός αυτός και ε, ε, ήξερα ότι υπήρχε δυνατότητα να χρηματοδοτήσει κανείς ε, ορισμένους τομείς αλλά εγώ γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι προτάσεις οι οποίες γίνονται και ε, βέβαια θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι χειρότερος κακοπληρωτής από τους υπολείπους για πολλούς και διάφορους λόγους τους οποίους μπορώ να αναφέρω. Μπορώ δηλαδή να σας πω γιατί είναι κακοπληρωτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτοί είναι πόδινοι λόγοι. Δηλαδή έχουν στενή σχέση με μία πολιτιστική αντιμετώπιση αποφυγής κινδύνων. Στον τομέα των εμπειρογνωμόνων και των υπευθύνων για τη λήψη των αποφάσεων. Υπάρχει μια σαφή στάση. Οι αποφάσεις σχετικά με τις πληρωμές είτε ε, σπρώχνονται προς τα πίσω είτε καθυστερούνται διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, κανόνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή ε, θα πρέπει όποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να μην κάνει κανένα λάθος. Ε, εάν λοιπόν δεν αλλάξει η κοσμοθεωρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ασχέτως όμως από αυτό το ψυχολογικό παράγοντα επέμεινα ότι θα πρέπει να προωθηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει ε, να μπορέσει να γίνεται σεβαστό, σεβαστή η αρχή της πληρωμής εντός 30 ημερών. Πρέπει να σας πω και για άλλους ε, λόγους ε, γιατί κινούμε προς αυτή την κατάφυση και γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ κακοπληρωτές δηλαδή υπάρχουν, ε, υπάρχουν ίσως καθυστερήσεις μέχρι και 10 χρόνια, είναι γνωστό αυτό. Εγώ διαπίστωσα ότι είμαστε ο χειρότερος πληρωτής διότι υπάρχει αποφυγή των ευθυνών και ούτω καθεξής. Ζήτησα όμως να λυθεί αυτό το πρόβλημα και θεώρησα ότι είναι ένα στοιχείο της αξιολογήσεως του προσωπικού μας. Δηλαδή ε, για τους γενικούς διευθυντές ζήτησα μέσα στην περιγραφή των καθηκόντων να αξιολογείται η ε, απόδοση ενός στελέχους και βάσει αυτού του στοιχείου. Και έτσι μπορέσαμε κάπως να προχωρήσουμε. Δηλαδή σήμερα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα και μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας πληρωμών. Δηλαδή τα πράγματα βελτιώνονται. Αλλά δεν θέλω να γενικεύω, δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ε, ανεκτό να θεωρούμε ε, ότι μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε στους άλλους τις δικές μας απόψεις χωρίς εμείς να σεβόμαστε οι ίδιοι. Και γι' αυτό ό,τι ισχύει για τους άλλους θα πρέπει να ισχύει και για μας. Ε, ε, Εύελιν, θα μπορούσα να σου διηγηθώ πολλές ιστορίες επί του θέματος αυτού στα πλαίσια του κοινωνικού δικαίου και θα σου εικονόταν η τρίχα στο κεφάλι. Δηλαδή υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις παραβιάσεων των ε, ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων που υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, τώρα, το άλλο θέμα που αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν αναφέρθηκα στο βασικό θέμα μας του πρώτου εξαμήνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι κάνουμε ό,τι είναι εφικτό. Είμαστε σε μία φάση τώρα όπου δεν χρειαζόμαστε δημιουργικότητα, επινοητικότητα, αλλά ακρίβεια στα πράγματα επί των οποίων έχουμε δεσμευτεί. Δηλαδή, εάν τα κράτη πράξουν αυτό το οποίο έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατήσουμε τις προθεσμίες τότε θα μπορέσουμε όντως να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πολύ καλύτερο πλαίσιο δραστηριότητος και αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο έχουμε αναλάβει να νομοθετήσουμε ε, και μπορώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία ελέγχθησαν εδώ. Δηλαδή, όσον αφορά την περαιτέρω ε, επέκταση της παγκομισμιοποίησης. Είναι σαφές ότι χρειάζεται μία ριζική αλλαγή των δομών των συγχρόνων βιομηχανιών οι οποίες γίνονται όλο και πιο παγκόσμιες, όλο και πιο διεθνείς. Είναι μία τάση που ενισχύεται συνέχεια και ε, θα υπάρχουν παραγωγές εκεί όπου είναι πιο προσοδοφόρες. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν σε ορισμένα σημεία χώροι εργασίας ε, στα περιθώρια της Ευρώπης και είναι μια τάση στην οποία ε, βλέπουμε να ενισχύεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις μας, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να απασχολήσουν και περισσότερο προσωπικό, όχι όμως υποχρεωτικά στην Ευρώπη. Και πρέπει να το δεχτούμε. Η όλη μας στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, να μην εξαντλήσουμε ε, τις ε, δυνατότητες αναπτύξεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην Ευρώπη για να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις επιχειρήσεις εδώ και θα επανόλθω στα αναφυγεία τα οποία ανέφερε η κυρία Σάλτερ Μόζερ. Εάν λοιπόν ε, συγκρίνουμε την Ευρώπη με την Αμερική βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές. Η Αμερική αναπτύσσεται πιο γρήγορα, ε, χρησιμοποιούνται πιο γρήγορα σύγχρονες τεχνολογίες. Είναι στοιχεία τα οποία έχουμε αναλύσει επακριβώς και έχουμε διατυπώσει όλες τις δυνατές και πιθανές προτάσεις και πιστεύω ότι για την διεθνή πολιτική δεν μπορώ να καταλάβω Πώ πως ένας πολιτικός λέγει όπως η κυρία Γκέπχαρτ ότι αυτό είναι το ουσιαστικό μας θέμα. Δεν πρόκειται για τις επιχειρήσεις ή για τους ιδιοκτήτες. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δεξαμενή ε, εργασία στην οποία έχουμε, να μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις εργασίας. Είναι ένα πολύ ζωτικό θέμα και πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Παραδείγματος χάρη πρέπει να δούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να λάβουν ευθύνες και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις. Είναι κάτι πολύ περίπλοκο, γι' αυτό και προσπαθούμε να μειώσουμε την ε, γραφειοκρατία. Συνεπάγεται όμως και ορισμένους κινδύνους, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να χρηματοδοτήσει κανείς μια επιχείρηση στην Ευρώπη από ότι στην Αμερική. Στην Αμερική αν είμαι νέος, Οπότε θα με χρηματοδοτήσει αλλά στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι έτσι ακόμη και αν πρόκειται για νέες ιδέες και υπάρχει όλο και περισσότερος δισταγμός του τραπεζικού συστήματος ο οποίος αποτελεί μια τροχοπέδη. Γι' αυτό θα αφήσω μία κληρονομιά στην Ευρώπη και ελπίζω ότι θα έχω πετύχει αυτό το οποίο συνειδητά επιζητώ, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όντως να μπορέσουν να είναι αποφασιστικές για το οικονομικό μας μέλλον και να μπορέσουν να λειτουργήσουν ε, απρόσκοπτα είναι ένα θέμα ε, το οποίο στηρίζω πλήρως. Ε, τώρα όμως έρχομαι στην κυρία Σάντερμόζερ. Κυρία Σάντερμόζερ, συμφωνώ από το Διαρθρωτικό Ευρωπαϊκό Ταμείο όταν μία επιχείρηση ε, ευρωπαϊκή καταρρεύσει δεν διατίθεται κανένας ε, ε, πόρος για να βοηθήσει το προσωπικό. Στο σύνολο, από πλευράς οικονομικής, Υπάρχει μία αλλαγή των δομών, βελτιώνεται η κατάσταση και οι θέσεις, που χάνονται, οι θέσεις εργασίας που χάνονται στον ένα τομέα μπορούν να αναπτυχθούν σε κάποιο άλλο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν στο ίδιο γεωγραφικό σημείο και την ίδια χρονική ε, στιγμή, στον ίδιο τομέα και χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες. Δηλαδή για τον εργαζόμενο σε ένα συγκεκριμένο σημείο είναι μια προσωπική καταστροφή. Είναι δηλαδή ε, κάτι το οποίο ε, εμείς ε, παραβλέπουμε όταν έχουμε μία μακροοικονομική αντιμετώπιση. Δηλαδή αυτό το οποίο παραβλέπουμε είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια προσωπικών δραμάτων και καταστροφών και υπάρχει μόνο ένα πράγμα Δηλαδή, δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε σαν ευρωβουλευτές ή σαν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει στην Ευρώπη για τους εργαζόμενους να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον ταχείας οικονομικής αλλαγής. Δηλαδή χρειαζόμαστε πιο ευρείες δεξιότητες, περισσότερες δεξιότητες, διότι ακόμη και στη χώρα σας Εάν δεν απατώμε, στη Δανία υπάρχει ένα θαυμάσιο πρότυπο για το πώς μπορεί κανείς να κάνει κάτι τέτοιο η ευελιξία από πλευράς των εργαζομένων για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους και για να δημιουργηθεί μία ασφάλεια κατά, εφόσον ε, θα μπορέσουν να υπάρξουν επιχειρήσεις που θα προσφέρουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή αυτή, αυτός είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επιβιώσουν της κρίσεως. Μόνο δηλαδή να τους βοηθήσουμε να αυξήσουν τις δυνατότητές, τις ικανότητές τους. Αλλά ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ή στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και στην ενδοεπιχειρησιακή δομή η οποία θα επιτρέπει αυτή την ευελιξία του εργαζομένου και θα τη διευκολύνει. Αυτή είναι η πείρα την οποία εγώ έχω αποκομίσει. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα ιδιορθρωτικά ταμεία. Είναι κάτι που δεν πρέπει να παραβλέψουμε, αλλά είναι ένα, πρόγραμμα, ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί μόνο του. Όταν, ε, όταν χρεοκοπεί ε, μία επιχείρηση λέγεται τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να συνεννοηθούμε. Δεν θα μου επιτρέπατε να χρησιμοποιήσω δημοσιονομικούς ευρωπαϊκούς πόρους και ε, να επέμβω σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είναι κάτι που δεν προβλέπεται από τους κανόνες μας. Αυτό δεν μπορούμε να το πράξουμε, αλλά για τον τομέα ο οποίος πλήττεται μπορούμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες πλαίσιο και θα δείτε παραδείγματος χάρη ότι ο ναυπηγικός τομέας ήταν ο πρώτος στον οποίο χρησιμοποίησαμε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή η πρωτοβουλία η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή αυτού του αιώνα και αυτής της δεκαετίας επέτρεψε να αντεπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό και είναι κάτι το οποίο έγινε τελείως συνειδητά. Δηλαδή ξέραμε ότι είναι ένας ευαίσθητος τομέας η ναυπηγική βιομηχανία υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες οι οποίες ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Οι Κινέζοι έχουν εκδιώξει ε, τους Κουβανούς ε, τους, ε, και τους Κορεάτες και τους Ιαπωνέζους από την αγορά αυτή. Θέλουν να υπερισχύσουν των Ευρωπαίων, θέλουν να δημιουργήσουν ειδικά είδη πλοίων και οι μόνες δυνατότητες που έχουν τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία είναι τεχνολογική πρωτοπορία όπου ε, κατασκευάζονται πλοία όπου το κόστος δεν είναι τόσο βασικός τομέας. Λοιπόν, ε, εγώ είμαι ε, πολύ, αφιβάλλω πάρα πολύ αν μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Κορέα διότι οι Κορεάτες αρνούνται να προβούν ε, και να ε, ασχοληθούν με διαιτησία στα πλαίσια του ΟΣΑ. Υπάρχουν ε, διάφορες πρακτικές οι οποίες εξασκούνται εις την Κορέα εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και έχει ασχοληθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει όταν ιδίως σκεφτόμαστε την κατάσταση των ευρωπαϊκών ε, ναυπηγείων και τα ναυπηγεία δεν είναι τα μόνα που μας απασχολούν. Την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη Βρέμη σε ένα συνέδριο για την ναυπηγική βιομηχανία όπου θα συνέλθουν πάρα πολλές χώρες και οι εμπλεκόμενες. Θα προσπαθούμε δηλαδή κάτι να κάνουμε από αυτού. Ε, Κυρία Ράπτη, δεν κατάλαβα τι εννοούσατε όταν μιλήσατε για τη φαρμακοβιομηχανία. Ε, αναφερθήκατε στα δικαιώματα των ασθενών και ε, στο δικαιώμα πληροφόρησης. Δεν ισχύει ότι δεν το ζήτησαν οι ασθενείς. Το ισχύον δίκαιο απαγορεύει να υπάρχει διαφήμιση και πληροφόρηση για τα φάρμακα που συνταγογραφούνται και όλο και περισσότερο προσπαθεί, ε, υπάρχει προσπάθεια να παρακαμφθεί αυτός ο κανένας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό προσπαθεί να ε, ενισχύσει την απαγόρευση διαφήμισης με το να διατυπώνει ε, σαφώς τα δικαιώματα πληροφόρησης των ασθενών για τα φάρμακα που συνταγογραφούνται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται οποιοδήποτε κερδίζει χρήματα δηλαδή ε, από την ε, από αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή όποιος τα παράγει, όποιος τα εμπορεύεται γνωρίζει τα πάντα για το φάρμακο αυτό και μόνο αυτός ο οποίος πρέπει να τα χρησιμοποιήσει δεν ξέρει τι συνεπάγεται η λήψη των φαρμάκων αυτών είναι τελείως ουτοπία να πιστέψουμε ότι δεν έχει δυνατότητα πληροφόρησης ο ασθενής παρόλο που και εκεί δεν υπάρχει ε, διαφήμιση αλλά όποιος έχει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μάθει τα πράγματα που χρειάζεται για ένα φάρμακο αυτό το οποίο δεν έχει ελεύθερα είναι την διαφήμιση και την πληροφόρηση είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ του τι επιτρέπεται και του τι όχι και γι' αυτό διατύπωσε αυτή την ε, πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό κατόπιν ε, προτάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ε, ακόμη και αν δεν το θε ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποχρεωθήκαμε να το πράξουμε διότι μας το ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Μάντερς, όσον αφορά την ευρωπαϊκή εναρμόνιση των συστημάτων συναγερμού. Δεν το γνωρίζω καλά αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για εναρμόνιση και του τι μπορούμε να κάνουμε στην ευρωπαϊκή εναρμόνιση και στην τυποποίηση ε, μέσω της Γενέβης και των σχετικών οργανισμών διότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κατασκευαστές. Εμάς μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε το θέμα από πλευράς περιβαλλοντολογικής ενδιαφέροντος και εκεί είναι ε, απαραίτητο και αυτά τα οποία κάναμε με τους ε, χάρτες παραδείγματο χάρη ε, ήταν κάτι το οποίο κάναμε για περιβαντολογικούς λόγους. Ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω κύριε Μάντερς ένα λεπτό να σκεφτείτε αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά το θέμα του track record, διότι ε, είμαι υπεύθυνος και για την έρευνα και με απασχολεί η έρευνα ιδίως όσοι έχει σχέση με την εσωτερική ασφάλεια με, για την τρομοκρατία και για τα εγκλήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι πρόκειται για θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και χρειάζονται πολύ χρόνο. Ξέρετε γιατί τα θέματα αυτά είναι πολιτικά ευαίσθητα risk of invading privacy. Δηλαδή κίνδυνος να επέμβει κανείς στην ιδιωτική ζωή. Μπορώ να σας πω τι τεχνικές υπάρχουν που διατίθενται αυτή τη στιγμή που επιτρέπουν τη δυνατότητα του person tracking να παρακολουθεί κανείς έναν ιδιώτη και να ξέρει ανα πάσα στιγμή που βρίσκεται ένα άτομο και τι κάνετε. Η τεχνολογία αυτή υπάρχει. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα, το car tracking. Πρέπει όμως να δούμε αν είναι κάτι το οποίο πραγματικά επιθυμούμε να έχουμε. Μισελ. Μισελ Μπαρνιέ, είναι ωραίο το ότι βρίσκεσαι και εδώ πάλι και συναντηθήκαμε. Λοιπόν, για τις ε, αντιρρήσεις για την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών είμαι πρόθυμος πιο εμβαθυμένα να έχω μια προσωπική συζήτηση μαζί σου. Δεν πιστεύω εγώ ότι αυτοί οι φόβοι, αυτές οι φοβίες θα υλοποιηθούν. Δεν πιστεύω για παράδειγμα ότι ο δημόσιος τομέας θα είναι επιφυλακτικός με παραγγελίες που θα, δινών, θα έδινε αν συγκεκριμένοι στόχοι πληρωμών πρέπει να τηρούνται. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Έχουμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεράστιες διαφορές Έχουμε αυτού του αριθμούς εδώ για να το πω αυτό. Μια στιγμή. Πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία, οι αριθμοί. Εδώ, έτσι, ωραία. Λοιπόν, να σα αναφέρω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Ακούστε. Λοιπόν, οι πραγματικές πληρωμές που γίνονται. Δέκα ημέρες τώρα για, τις, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τροποποίηση του νομικού πλαισίου πρόσφατα. 15 μέρες Φινλανδία, Ιρλανδία, 30 Λουξεμβούργο και Σουηδία, 45 ημέρες στη Γαλλία, 60 στην Ισπανία, 90 στην Ιταλία και μετά Ελλάδα, πέρα από, πέρα από <laughs> τα όρια του καλού και του κακού. Τώρα, είναι δυνατόν και πολλά παραδείγματα το δείχνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πληρωμών χωρίς να απεμπολίσει το κράτος ε, τη δυνατότητα σύναψης ε, παραγγελιών και συμβάσεων. Δεν νομίζω λοιπόν θα υπάρξει ένα τέτοιο πρόβλημα. Είπα, αυτό που αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, νοσοκομεία και άλλα τέτοια κοινωνικά θεσμικά όργανα, η πρότασή μας προβλέπει σίγουρα την δυνατότητα εθνικές ε, εξαιρέσεις να ισχύσουν. Αλλά είμαι πρόθυμος να το ξανασυζητήσω αυτό σε αυτή την πτυχή του. Τώρα, το άλλο θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμιευτηρίου. Αυτό είναι, θα έλεγα, ένα θέμα το οποίο δεν αφορά το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Θα έπρεπε, συνάδελφος, να τοποθετηθεί. Έχω μεγάλη συμπάθεια για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ως μόνο στόχο τους των συναλλαγών τους τη μεγιστοποίηση των κερδών. Εγώ προέρχομαι από την Γερμανία που έχει τελείως διαφορετική δομή η δομή των τραπεζών από τις άλλες χώρες όπου έχουμε δημόσιες ε, κρατικές τράπεζες με ένα συγκεκριμένο στόχο και έχουμε συνεταιριστικές τράπεζες, ταμιευτήρια δηλαδή με τομεακή δραστηριότητα. Δύο τρίτα λοιπόν ε, ε, αυτών των ιδρυμάτων στη Γερμανία δεν εντάσσονται, δεν υπάγονται στη μεγιστοποίηση των κερδών ως αρχή. Πολλές φορές έχουν υπάρξει αντιρρήσεις όσον αφορά τους γκουρού των οικονομικών, ιδιαίτερα όσον αφορά το Λονδίνο. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, ε, καταδείχθηκε ότι αυτό ήταν κάτι το πολύ χρήσιμο ως θεσμός για μας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για ένα ευρύτατο πλαίσιο σχολείων. Να ξαναδούμε τώρα τα θέματα αυτά. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ξεπεράσει κάπως το χρόνο μας, ο οποίος πιέζει. Η κυρία Ράπτη ζητεί τον λόγο. Α, θα ήθελα να δω να ζητήσω αν είναι δυνατόν σε σχέση με τις ερωτήσεις για ένα τέταρτο. Πέντε έχω που ζητούν να παρέμβουν. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, να ζητήσω χωρίς να θέλω να αναστείλετε την δημιουργική σας δραστηριότητα. να σας σε συντομότατη. Σβάμπ, Στήλερ, Μάλερ, Βιουβάν και Κέλλη. Λοιπόν, το, το τελευταίο λεπτό εσείς και η κυρία Ράπτη θέλει να επανέλθει αλλά νομίζω αν μπορείτε στον κύριο Φεχόγεν ε, ε να συζητήσετε μαζί του υστερότερα. Οι πέντε αυτοί συνάδελφοι λοιπόν ζητώ να είναι συντομότατοι στα σχόλιά τους για να δώσουμε ευκαιρία στον κύριο Φεχόγεν να ολοκληρώσει και θα τελειώσουμε στις πέντε παρατέτατο. Ο κύριος Σβάμπ, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ που τόσο γοργά ήρθατε και πάλι στην Ευρωβουλή μετά τις εκλογές. Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει η προεργασία και πριν από τις θερινές διακοπές. Τώρα αυτή η εργασία για τους επόμενους μήνες θα είναι ιδιαίτερα θελκτική για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την προεργασία σα. Θα ήθελα όσον αφορά την οδηγία για πληρωμές να μην πω τίποτα. για τις θέσεις πληρωμών έχουν αναφερθεί αρκετά θέματα. Εδώ στο σχέση με το Small Business Act να αναφέρω κάτι. Σίγουρα είναι πολύ θετικό ότι η δημόσια προσοχή στρέφεται σε αυτό το πρόβλημα και που έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση ε, για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά τη θητεία σα, αλλά κυρίω ψυχολογικά ζητήματα ή στοιχεία εντάσσονται εδώ που διαδραματίζουν ένα ρόλο, μεγάλο ρόλο και καταφέρατε να ε, τύχει μεγαλύτερης προσοχής σε αυτό το θέμα. Τώρα, αν στο τέλος ε, τα επιμέρους μέτρα θα συμβάλλουν, θα συνεισφέρουν ε, για την επίρρευση του τελικού στόχου, δεν εξαρτάται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωβουλή, αλλά και την αντιμετώπιση των επιμέρους εμπλεκομένων. Και φυσικά θα πρόκειται για το θέμα και εσείς με το παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αξιολόγηση των υπαλλήλων σας ε, όσον αφορά την δυνατότητα υλοποίηση διαφορετικών δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, πόσο γοργά δρά η πολιτική, πόσο γοργά αντιδρούμε εμείς. Και ιδιαίτερα στον τομέα της γραφειοκρατίας που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερη επιβάρυνση, διαπιστώνουμε ότι σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία εσεί εισαγάγατε και αναφερθήκατε σε αυτά, χαίρομαι που τα ε, θυμόσαστε εσείς ε, το θέμα τώρα το οποίο εσείς ε, συνδέσατε με, την δική, με το δικό μου άτομο την δραστηριότητά μου θέματα για παράδειγμα που προσπαθούν ευρωβουλευτέ, ευρωβουλευτές όπως και εγώ να θέσουμε στο προσκήνιο κράτησε τρία χρόνια μέχρι ότου να καταλήξουμε σε επιβολή διεθνών προδιαγραφών και όχι μόνο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτό δεν είναι επίκριση αλλά θα έπρεπε να λάβουμε επίσης υπόψη να εξετάσουμε ποιες δυνατότητες επιτά επιτάχυνση έχουμε, ποιες δυνατότητες έχουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε τέτοια, τέτοιου είδους θέματα στο μέλλον πιο γοργά να μπορούν να διευθετούνται. Ευχαριστώ. Um, uh, ε, Στήλερ, την οποία τη βλέπουμε μετά από πολύ καιρό. Χαιρόμαστε όλες, ε, όλος ιδιαίτερος ε, που επανήλθατε. Ευχαριστώ πολύ, Μάλκολ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο ε, αφορά τις μικρές επιχειρήσεις και την ε, ε, και τις θέσεις απασχόλησης. Μιλήσατε για τη δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης, μας δώσατε και κάποια στοιχεία αριθμητικά Μιλήσατε για τεράστια ποσά που δόθηκαν ε, στις μικρές επιχειρήσεις ε, και μάλιστα και υπάρχει και ένα σχετικό άρθρο, το ε, Stopping Startups, στον αμερικανικό τύπο για το θέμα αυτό. Ε, μπορούμε να το δούμε αυτό μέσω του Facebook, μέσω του Google, ε, μέσω του Yahoo. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ ε, άμεσα. Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα το θέμα των επιχειρήσεων startup γιατί έχουμε μικρό χρόνο, λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Παρόλα αυτά, επειδή θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί και επειδή μιλάμε για ε, κάποιες αρχές ε, οι οποίες είναι πολύ ικανοποιημένε με, το 30, με τις 30 ημέρες αλλά έχουν κάποιο πρόβλημα με το 5% που προτείνεται. Γι' αυτό προτείνω... Ε, Επειδή κάποιες τοπικές επιχειρήσεις ε, έχουν, κάποιες τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν γρηγορότερα σε αυτό, πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ειδικότερα αυτήν την πρωτοβουλία, να προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε κάτι τέτοιο, να μην υπάρχει δηλαδή αυτό το 5% το οποίο δεν ε, εξυπηρετεί το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε ε, για τις καθυστερημένες πληρωμές γιατί ούτως ή άλλως δεν ε, πρόκειται για καθυστερήσεις που προκύπτουν κυρίως από τις τοπικές αρχές, πρόκειται για καθυστερήσεις που προκύπτουν από άλλου είδους επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μπάρμπαρα Βάιλερ. Ναι κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με την οδηγία για τις καθυστέρησεις πληρωμών late payments. Διάβασα ότι αυτά τα 86 δισεκατομμύρια που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στη Γερμανία 50 δισεκατομμύρια είναι. Λέει ο μιλήτρια 50 εκατομμύρια, 50 δις. Είναι πολύ ανώτερο λέει το ποσό. Πολύ ανώτερο λέτε. Ναι, γιατί διαφορετικά θα είχαμε πάνω από το ίμιση. Εμείς έτσι δεν είναι. Και αυτό θα ήταν κάτι, θα έλεγα, εξωπραγματικό. Θα ήθελα να μου πείτε, εν τω μεταξύ έχουμε μια ολόκληρη σειρά σχολείων από ενώσεις και συλλόγους που ακούσαμε, από τις πιο ε, διαφορετικές ενώσεις και συλλόγους. Και είναι σημαντικό τι λένε οι εκπρόσωποι των Δήμων και κοινοτήτων. Θα ήθελα να ξέρω πιο πριν, αγαπητέ Γκούρτε Φεχόγερ, τι γίνεται, πώς πιο πριν οι τοπικοί εκπρόσωποι οι Δήμοι και οι κοινότητε αντέδρασαν, το χαιρέτησαν αυτό ως μέτρο ή ποια ήταν η αντιμετώπιση τους σε αυτό. Διότι επιπλέον άκουσα ένα ακόμα χειρότερο αριθμητικό στοιχείο το ότι ένα μεγάλο, μια μεγάλη πλειοψηφία των επιμέρους αυτών δεν μπορούν καν να ανακτηθούν αυτά τα ποσά, αλλά χάνονται. Είναι μια απώλεια που φυσικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική, ιδιαίτερα μειονεκτική θα έλεγα. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Το δεύτερο τώρα στις ε, θεμελιώδεις ε, τοποθετήσεις σας για ενισχύσεις ή επιδοτήσεις. Είπατε δεν επιτρέπονται ενισχύσεις ή επιδοτήσεις. Όλα τα άλλα θα πρέπει να είναι εξαιρεσει που τεκμηριωμένα θα πρέπει να εγκρίνονται ή όχι. Και εγώ θα ήθελα εδώ να πω, ε, εντάξει, όχι εθνικές εξαιρέσεις. Να πει κανείς για Ιταλικά ή Γερμανικά αυτοκίνητα θα υπάρχει κάποια εξαίρεση γιατί αυτά πρέπει να προστατεύονται, όλα τα άλλα δεν αξίζουν, δεν χρειάζεται να προστατευτούν. Όχι. Κάτι τέτοιο δεν αποβαίνει προ ε, όφελο των δικών μα στόχων. Δεν πρέπει να υπάρχουν ε, ειδικέ εθνικέ εξαιρέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμω να υπάρχει και κοινωνική συνένεση. Και νομίζω ότι αυτό στη σημερινή συγκυρία είναι σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν περιπτώσει όπου πραγματικά γίνεται προσπάθεια και από ε, εργαζόμενους την κακή διαχείριση των προηγούμενων ιδιοκτητών να την αντισταθμίσουν, να ενταχθούν εκείνοι και να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση η οποία θα έχει θετικές προοπτικές. Δεν πρέπει να χάσουμε το θετικό με το αρνητικό το οποίο θέλουμε να απαλείψουμε, να ρίξουμε δηλαδή τα νερά από, από την πανιέρα του μωρού και να πετάξουμε και το νερό στον υπόνομο εδώ θα πρέπει να δούμε και το θέμα της αντιμετώπισης της ε, μη χρηστής διαχείρισης. Ε, πρέπει να δούμε ίσως ε, το πώς θα μπορούσαμε θετικά να δράσουμε. Ίσως σε ένα κοντινό μέλλον να έχουμε μια νέα δυνατότητα αξιολόγησης ή εκτίμησης των επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Διότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε κάτι τέτοιο να λειτουργήσει. Υπό την παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της διεθνούς παγκόσμιας κρίσης. Τώρα, σε σχέση με τους γεωργικούς ελκυστήρες για τα τρακτέρ, δεν χρειάζεται να πω τίποτα και εγώ παραπάνω. Αληθεύει ότι και εγώ είχα εμπλακεί, όμως για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια εδώ, θυμάμαι και πρέπει να το πω αυτό, θυμάμαι ότι ένα μεγάλο μέρος της ενοχής δεν ήταν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε και των χριστιανοδημοκρατών του κ. Σβάμπ, αλλά οφειλόταν στην Ένωση των Παραγωγών Τρακτέρ, Γεωργικών Ελκυστήρων, που δεν είχαν πνεύμα θετικής, ε, θετικής συνεργασίας ε, και πρέπει να το πούμε αυτό. Χρειάζεται για την λειτουργία και εφαρμογή ε, προτύπων ε, και προδιαγραφών ασφάλειας ε, μια ενιαία τοποθέτηση των ενώσεων παραγωγών. Δεν το κάνανε τότε αυτοί. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες αρνηθήκαμε να εγκρίνουμε μια ξεχωριστή πορεία και τώρα το ξανά έχουμε το θέμα μπροστά μας. Τελευταίο σημείο, κρίμα επίτροπε που δεν μας το είπατε πιο πριν, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τηρεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες και είναι κακοπληρωτής. Κρίμα, <laughs> διότι για μένα αυτό είναι ακριβώς ε, εξίσου θα έλεγα καινούριο ενοχλητικό όπως και για σας. Αν θα το γνώριζα αυτό θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει σε μια διαδικασία προσφυγής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΚ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το κάνουμε αυτό και ούτως ή άλλως. Ε, και μπορείτε να βασιστείτε ότι αυτό σίγουρα θα πρέπει να είναι ένα θέμα για να δούμε πώς οι νέοι επίτροποι θα, είναι, θα αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα, δηλαδή τήρηση οδηγιών που έχουν εγκριθεί από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουβάν. Ο κύριος Ζουβάν παρακαλώ. Mm. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας που ήταν πάρα πολύ σαφής. Μιλήσατε κυρίως για την αναγκαιότητα μιας καλύτερης ρύθμισης, πιο εφιούς, πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ε, συμπολιτών μας και νομίζω ότι οι εξελίξεις έχουν δείξει ε, αυτήν την ε, αυτή την ανάγκη των ε, πολιτών ε, να ανταποκρίνεται καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανάγκες τους. Ε, αναφερθήκατε στη χρήση όλων των ε, περιθωρίων ελιγμών που έχουμε, για παράδειγμα τη χρήση του σχεδίου οδηγίας ε, για την καθυστέρηση των πληρωμών ε, και είπατε ότι έτσι βελτιστοποιούμε τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Εμείς βεβαίως μόνο υπέρ ενός τέτοιου εγχειρήματος μπορούμε να είμαστε. Βέβαια, οι ιδιαιτερότητες του ε, στόχου αυτού θα συζητηθούν ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η καλύτερη λοιπόν νομοθεσία η οποία βελτιώνει σε το μέγιστο βαθμό ε, την εσωτερική αγορά έχει να κάνει με την εδραίωση ε, της, για, παρά, παράδειγμα της προστασίας της εσωτερικής αγοράς γιατί εντός εσωτερικής αγοράς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποφέρουν ε, από έλλειψη ισότητας και το αναφέρω αυτό σε σχέση με τον ανταγωνισμό ε, μεταποιημένων προϊόντων ε, από περιοχές που δεν έχουν τις ίδιες, τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα, ας πούμε, τις ίδιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ε, απολύτως ε, με αυτό που είπατε σε σχέση με την αναγκαιότητα βελτίωσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό της εσωτερικής αγοράς, της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ε, δεν διαφωνώ με όλους τους μηχανισμούς που αναφέρατε, ότι πρέπει να αναπτυχθούν, ότι πρέπει να τους εφαρμόσουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και άκρος ικανοποιητικό ε, το πρόγραμμα ε, που μας εξαγγείλατε, αλλά πρέπει να ε, δούμε ε, και την, πώς θα συνδυάσουμε τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αλλά και την εδραίωση των μέσων που έχουμε ήδη στη διάθεσή, σας, όπως, στη διάθεσή μας όπως είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εσάς να σας καλωσορίσω γιατί είστε νέο μέλλον της Επιτροπής μας, ο κύριος Κέλλη από την Ιρλανδία. Δύο παρατηρήσεις. Θα, είμαστε, θα είμαι σύντομο ε, στην Ιρλανδία, όπως και σε πολλές άλλες ε, χώρες, ε, γιατί εγώ προέρχομαι από τον τομέα μεταποίησης, που επλήγει πάρα πολύ από την κρίση και είναι καλό λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία να φτάνουν καλά ευρωπαϊκά νέα για τους λόγους που φαντάζεστε. Το Ταμείο για την Προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση ε, ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο ε, στην Ιρλανδία, όπως επίσης και το πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στους τομείς που κυρίως επλήγησαν, όπως για παράδειγμα ο μεταποιητικός τομέας. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κρίση και η έλλειψη άμεση άμεσης ανταπόκρισης στους κινδύνους είναι κάτι το οποίο ε, μας δημιουργεί κάποια ανησυχία και κάποια σύγχυση μπορώ να πω. το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτό εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και αναφέρομαι κυρίως στην τεχνολογία που αποτελεί την υποδομή ε, του τομέα της ενέργειας. Θα μπορούσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όσον αφορά την, ε, ε, την, τεχνολογία που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε για παράδειγμα υψηλές προδιαγραφές για να μπορούμε να είμαστε και, να μπορούμε, να είμαστε και δημιουργικοί, παραμένουμε δημιουργικοί. Και θα ήθελα να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο για την, για την οδηγία περί καθυστέρησης ε, πληρωμών. Εμείς το γνωρίζουμε, τη γνωρίζουμε αυτή την κατάσταση στην Ιρλανδία και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουμε αφήσει απ' έξω, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τομείς συγχρηματοδότηση ε, με φιλανθρωπικές οργανώσεις κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ε, γιατί ε, δίνουμε τόσο ιδιαίτερη σημασία στον ιδιωτικό τομέα, μπορούμε να, δώσουμε, να δώσω πάρα πολλά παραδείγματα όπου υπάρχουν πολύ σοβαρές ε, απώλειες θέσεων εργασίας γιατί ακριβώς ε, δεν έγιναν σεβαστές κάποιες προδιαγραφές και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε στους επίμονους παραβάτες κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν κάνουμε επαρκώς. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όλα αυτά τα οποία μας είπατε ε, σε γενικές γραμμές μας βρίσκουν σύμφωνους και θα συμμετέχουμε στον αγώνα για να τα πετύχουμε. Ο κύριος Φεχόγεν, πολύ σύντομα παρακαλεί ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία αυτή με τους γεωργικούς ελκυστήρες στα τρακτέρ ολοκληρώνεται τώρα ε, και τη νέα οδηγία θα σας την παρουσιάσω όταν θα είναι στη διάθεσή μας. Αν είναι πραγματικά μια ατυχής ιστορία θα έλεγα, μια ε, ε, βεβαρημένη ιστορία. Και ευχαριστώ την κυρία Βάρη, τον κύριο Σουβάμπα. Και πρέπει να πω ότι δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη πίεσης ε, και υπαναχώρηση και έτσι λοιπόν προχώρησε το θέμα. Για την κυρία Στήλερ να πω ότι η έννοια που χρησιμοποίησε exchange of good practices, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και το να μάθει ο ένας από τον άλλον. Στον τομέα της, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει απόλυτα κεντρική σημασία, θεμελιώδη σημασία και αυτό είναι μια κυριότητα τη δραστηριότητά μας ε, σε σχέση με τις, ε, τα κρατημέλη και τις επιχειρήσεις, με την ανταλλαγή αυτών των, βέλτιστων πρακτικών και ανταλλαγή ε, πείρας ε, να έχουμε την προαγωγή των επιχειρήσεων μεταξύ τους αλλά και την προσέγγιση των κρατικών υπηρεσιών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το πλαίσιο. Είμαι πρόθυμος να σας διαθέσω τεκμηριωμένο κατά υλικό γι' αυτό και το μεγαλύτερο business support δίκτυο παγκόσμια αυτό που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος τέλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικτύωση γνώσεων και πείρας που στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουμε στη διάθεσή μας και που θέλουμε να προαγάγουμε. Έχουμε μια εξαιρετική πείρα εδώ, εξαιρετική εμπειρία και μπορούμε να δούμε σαφέστατα πώς οι ιδέες που αναπτύχθηκαν σε μια χώρα διαχέονται και ξαφνικά σε άλλες χώρες υιοθετούνται. Εμφανίζονται κάποια πράγματα που καταρχήν στη Δανία ίσως υιοθετούνται και μετά ξαφνικά στην Πορτογαλία συνεχίζονται. Πράγματα που κάποτε ξεκίνησαν στο Λουξεμβούργο ξαφνικά εμφανίζονται στη Βουλγαρία και τα λοιπά. Τα είδαμε όλα αυτά και τα ζήσαμε και είναι ωραίο να το ζει κανείς κάτι τέτοιο, να το βιώνει αυτό. Αλλά σίγουρα συμφωνώ ότι είναι θεμελιώδους σημασία στοιχείο αυτό. Τώρα, για τον συνάδελφο στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, προσέξτε, ή τουλάχιστον όσον αφορά του ανταγωνιστέ του στι παγκόσμιε αγορέ, στι διεθνεί αγορέ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο να εκτίθενται την παγκόσμια ανταγωνιστική τάση, η περιβάλλον. Είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο αυτό. Εκείνε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη που ασχολούνται με παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο είναι σε υψηλό βαθμό εξειδικευμένε. Παράγουν ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο προϊόν για το οποίο είναι ανταγωνιστικές και ε, σε παγκόσμιο πλαίσιο παρότι δεν μπορεί να είναι οι μόνες. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν έχει, α το πω έτσι και απλά, μία πτυχή που συναντάται και με το μέγεθος των επιχειρήσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκείνες που υιοθετούμε εμείς ε, υπό τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι πολύ μικρές για να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Και γι' αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν βρίσκονται εκτεθειμένες σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, αλλά στον ευρωπαϊκό. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες δυνατότητες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποιοι φραγμοί, κάποια εμπόδια που είναι αναπόφευκτα. Ας μην αυταπατώμαστε. Η πολυ ποικιλομορφία της ε, πολιτισμικής μας παράδοσης για την οποία είμαστε περήφανοι στην Ευρώπη είχε ένα μειονέκτημα εδώ για μας στις ΗΠΑ, στην Αμερική, φτάνει μια γλώσσα όλοι και όλοι για μια επιχείρηση. Παντού με τα αγγλικά συνεννοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε εμάς όχι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στη Λιθουανία έχει πρόβλημα. Αν θέλει παντού στην Ευρώπη να είναι, προσβα... Ε, να είναι διαθέσιμα τα προϊόντα της στη γλώσσα της. Αντιμετωπίζει πρόβλημα λοιπόν, γλωσσικό πρόβλημα, πολιτισμικής ποικιλομορφία πρόβλημα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιβαρύνονται και δυσχεραίνονται στο έργο τους από αυτή την ποικιλομορφία σίγουρα. Όμως το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη και το συνυπολογίζουμε. Αυτού του είδους οι φραγμοί, οι πολιτισμικοί και άλλοι παρόμοιοι συναφείς μπορούν να απαλληφθούν ή να συρρυκνωθούν, να μειωθούν. Τώρα για τις εισαγωγές. Εισαγωγές από χώρες που έχουν μικρότερο κόστος παραγωγής και όσον αφορά κοινωνικές παροχές ε, η προστασία του περιβάλλοντος ε, υιοθετούν ένα dumping και γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι στρεβλή διαδικασία και ε, πρέπει να καταπολεμηθεί. Παντού όπου υπάρχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή άλλες προδιαγραφές ισχύουν για εκείνους που εξάγουν σε εμά οι ίδιοι κανόνες, οι, ίδιοι, λοιπόν, οι ίδιες προδιαγραφές. Κάποιος που από την Κορέα ή την Ιαπωνία ή από αλλού θέλουν να, εισάγουν, να εξαγάγουν κάτι σε εμά για να εισαχθεί σε εμά, ε, το, το προϊόν του πρέπει να ανταποκρίνεται στι δικέ μα προδιαγραφέ. Είναι σαφέ αυτό. Και αυτό τώρα όσον αφορά για την Κίνα έχουμε μια άλλη όψη του ε, νομίσματος Πολλές χώρες ε, παγκόσμια έχουν ε, μικρότερο κόστος παραγωγής και λαμβάνουν λιγότερο υπόψη την προστασία του ε, περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας ή της οικολογίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεταβαίνουν επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες και παράγουν αλλού με μικρότερο κόστος παραγωγής. Και στην Ευρώπη εστιαζόμαστε στην υψηλότερη ποιότητα και τεχνολογία εχμής. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πρότυπο ή αν πρέπει να αλλάξει. Αλλά σε ένα σημείο πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρέπει να ε, εργαστούμε με ιδιαίτερη ένταση και να ασκήσουμε πίεση εμείς ως Ευρωπαίοι, ώστε είτε μέσω διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, είτε μέσω ε, εθελοντικών κωδίκων ε, δεοντολογίας, οι προδιαγραφές για την κοινωνία, κοινωνική συνιστόσα και το περιβάλλον να μπορέσουν να αναβαθμιστούν στις χώρες αυτές θα ήθελα οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, να υιοθετήσουν ένα διοντολογικό κώδικα που θα τις υποχρεώνει, θα τις αυτοϋποχρεώνει στις χώρες που παράγουν εκτός Ευρώπης και από τις οποίες εισάγουν να εφαρμόζουν τις ίδιες προδιαγραφές που εφαρμόζουν στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, να υποχρεωθούν αυτές οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις και το πρόβλημα θα έχει άλλες διαστάσεις. Κύριε Κέλλη, ευχαρίστω σημειώνω αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε. Και σίγουρα στο έργο μας θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας και ούτω ή άλλω για τι συγκεκριμένε δραστηριότητε και πρωτοβουλίε εντάσσονται σε σχέση με τι αρμοδιότητε τη δική σα κοινοβουλευτική επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο και θα ξανάρθουμε ω Επιτροπή σε εσά και θα σα αναφέρουμε τα σχετικά. Στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία πρέπει κάποια πράγματα να αναθεωρηθούν και να τα ξαναδούμε. Θα πρέπει να ξαναδούμε στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία πώ θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αφενό κάποιε συγκεκριμένε βιομηχανίε τι οποίε χρειαζόμαστε ώστε η οικονομία μας να μπορεί να είναι αηφόρα και ανταγωνιστική, να μπορέσουν να διατηρηθούν στην Ευρώπη, με έδρα την Ευρώπη. Και θα πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα, ποιες τεχνολογίες πρέπει να κατέχουμε στην Ευρώπη εμείς και ποιες τεχνολογίες εμείς οι ίδιοι πρέπει να εφαρμόζουμε και να χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη και να δούμε ποιες επιπτώσεις θα συναχθούν από αυτές τις απαντήσεις. Παράδειγμα, αυτές τις τεχνολογίες χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, με αυτές τις τεχνολογίες πρέπει να, παράξουμε, να παράγουμε στην Ευρώπη και τι θα γίνει αν υπάρξει αλλαγή της κατάστασης με συνιστώσεις που προανέφερα πιο πριν, ε, με την κατάσταση επιχειρήσεων εξωευρωπαϊκά κτλ. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να καλυφθούν. Και στο τέλος, εδώ πρέπει να να ε, διορθώσω κάτι, να επανορθώσω Μάκομ. Είχατε δίκιο να διαμφισβητήσετε το ποσό το οποίο ανέφερα. Κατέληξα στην λάθος γραμμή. Θα σας δώσω δύο αριθμητικά στοιχεία. Όμως είναι εγγυημένα αυτά αυτή τη φορά, εντάξει. Το πρώτο αριθμητικό στοιχείο είναι ο συνολικός όγκος των δημόσιων παραγγελιών και συμβάσεων, public procurements στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι άκουσον άκουσον 1943 εκατομμύρια, δηλαδή 1,9 δις. Δηλαδή αγγλικά trillions, εντάξει, συνεννοούμαστε. 3 εκατομμύρια. Στη, στα γερμανικά μπιλιόνεν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μπιλιόνεν και τριλιόνεν. Με η αντιστοίχηση από τη μία γλώσσα στην άλλη δίνει άλλα ποσά. Τουλάχιστον πάρα πολύ μεγάλος όγκος χρημάτων είναι αυτός εντάξει. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Τώρα όμως και τώρα το επόμενο αριθμητικό μέγεθος, το επόμενο στοιχείο. Αν το καταφέρουμε τελικά και το πετύχουμε, οι, ο δημόσιος, οι δημόσιες παραγγελίες τον στόχο των 30 ημερών για εξόφληση λογαριασμών να τον τηρήσουν, τότε θα δημιουργήσουμε πρόσθετη φερεγγιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, άκουσον, άκουσον, 179 δις, 179 δις, λέει ο κύριος Φερχόγεν, 179 δις ευρώ. Εντάξει. Αυτή τη, αυτή τη φορά 179 billions Λοιπόν, μακροοικονομικά αυτά τα μεγέθη είναι τεράστια σημασία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Well, thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν άξιζε τον κόπο να καθυστερήσουμε λιγάκι και να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις. Ε, οι συνάδελφοί σα που έχουν κάνει τη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου θα έρθουν ε, να ε, μας δουν αύριο, οπότε θα μας πούν και εκείνοι και άλλα αριθμητικά στοιχεία, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κλπ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Uh, now, ladies and gentlemen, um, uh, we're running a bit late. Uh, Έχουμε λίγο καθυστερήσει, κυρίες και κύριοι. Και δεν θέλω να σας στερήσω τη δυνατότητα να πάτε στους, ε, να, πιείτε κάτι με τους Σουηδούς υπουργού, αλλά έχουμε και μερικά ακόμη θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκεκριμένα του κυρίου Μπούσόη. Οπότε όσοι αποχωρούν παρακαλώ να το κάνουν ήσυχα. Θα ήθελα να κάνω μερικές σύντομες ανακοινώσεις. Καταρχάς πρέπει επισήμως να εγκρίνουμε θα έπρεπε να εγκρίνουμε επισήμως τα πρακτικά της ε, συστατικής μας ε, συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου που βρίσκονται στο φάκελό σας, οπότε μπορώ να περάσω στην έγκριση των πρακτικών αυτών. Νομίζω περισσότεροι εξημών ε, είχατε παραβρεθεί. Επίσης, συμφωνήσαμε να έχουμε μία επιπλέον συνεδρίαση στις 7 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα, γιατί η Σουηδική Προεδρία μας ζήτησε να ε, έρθει να μας ενημερώσει για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα λάβει η χώρα στις 4 ε, Δεκεμβρίου. Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω επισήμως ε, να εγκρίνετε Ορισμένα ζητήματα για τα οποία είχε εργαστεί η προηγούμενη ε, Επιτροπή, στην προηγούμενη θητεία της και πρέπει να τα εγκρίνουμε ε, επισήμως και πάλι. Δικαιώματα των καταναλωτών πρώτη ανάγνωση. Ε, δεύτερον, το θέμα που έθεσε ο κύριος ε, Φερχόγεν για την καθυστέρηση των πληρωμών και ε, το θέμα των, της κλωστοϊφαντουργίας και των... Ε, την, την, την ε, ετικετοθεσία των ε, σχετικών προϊόντων. Θα ήθελα να σας πω ότι επισήμως θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας για τα θέματα αυτά τα οποία ανέφερα. Φυσικά, Πρόεδρε, δεν θέλω εδώ να δημιουργήσω ένταση. Όμω το δικό μου ημερολόγιο έχω καταχωρήσει και πιθανότατα όλοι στην αριστερή πτέρυγα. στι 7 Δεκεμβρίου θα έχουμε τη μεγάλη ευρωπαϊκή, το μεγάλο ευρωπαϊκό συνέδριο όπου κανονικά όλοι οι Ευρωπαίοι βουλευτές σε ε, αυτή τη νέα ε, ομάδα θα πρέπει να συμμετάσχουν. Έτσι, στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα αυτή. Απλά να το επαληθεύσουμε αυτό ακριβώς για την ημερομηνία, το ξαναδούμε. Κοιτάξτε, μία πρόταση έκανα. Αν θέλετε, ευχαρίστω να το αναθεωρήσω, να το συζητήσω και με τη Σουηδική Προεδρία. Θα επανέλθουμε για το θέμα αυτό στου συντονιστέ τότε. Απλώ ήθελα να σα το πω. Ανέφερα επίσης ε, κάποια στιγμή προηγουμένως ε, ότι σήμερα το πρωί κάναμε μια πολύ επί οικοδομητική συνάντηση με τους συντονιστές. Δεν θέλω να ε, σας ενημερώσω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορέσουμε να συζητήσουμε κυρίως για τα στρατηγική σημασία θέματα που συζητήσαμε με τους συντονιστές. Αυτό που αποφασίσαμε είναι να γίνει μια μεγάλη ε, και ευρεία συζήτηση ε, με τους συντονιστές οι οποίοι θα σας ενημερώσουν για τα θέματα αυτά. Θα συζητήσουμε κυρίως το θέμα της ανάθεσης των διαφόρων εκθέσεων και των μελετών ορισμένων ζητημάτων ε, που ε, πρόκειται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα γίνει λοιπόν μία συνεδρίαση 14 Σεπτεμβρίου για τους συντονιστές, αλλά ήθελα να λάβετε γνώση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής ε, πιστεύω θα ανατεθούν ε, ε, οι εκθέσεις στους συζητητές και στους σκιώδεις συζητητές. Σήμερα επίσης το πρωί συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που βρίσκονται εν εξελίξη, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεισφέρετε, θα ήθελα να μάθω πόσοι από εσά ενδιαφέρονται για τις ε, διάφορες εκθέσεις. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να σας πω. Το δεύτερο που ήθελα να ε, πω είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και πάλι να εξετάσουμε. Θα στείλουμε έξι μέλη της, της Επιτροπής μας ε, στη Σουηδία στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στη Στοκχόλμη και οι συντονιστές ε, των ε, ε, ομάδων πρέπει να ορίσουν μέλη για την αποστολή αυτή, για την ομάδα που θα επισκεφθεί την Σουηδία. Για ορισμένα στρατηγικά ζητήματα θα γίνουν συζητήσεις. Αυτά ήθελα μόνο να σας πω Ω ανακοινώσει του Προέδρου και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη, που είναι ο προπολογισμό 2010. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης και των τροπολογιών. Ο κύριος Νιούτον Ντάν ε, έφυγε και ο κύριος Μπουσόη ανέλαβε τα ε, καθήκοντα, ε, τα σχετικά καθήκοντα, υπέβαλε τη σχετική έκθεση και θα την ψηφίσουμε αύριο αφού ακούσουμε τον Σουηδό Υπουργό. Νομίζω ότι και ο κύριος Μέιορ από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ είναι εδώ, θα μας πει και την άποψη της Επιτροπής για το θέμα αυτό και όποιος ε, άλλος θέλει να παρέμβει, ε, ευχαρίστως. Κρίστιαν Μπουζόη, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ για πόση ώρα για όσο λιγότερο γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να κάνω μερικά σχόλια γενικά και μετά να είμαι λίγο πιο λεπτομερή όσον αφορά τι τροπολογίε. Σε σχέση με το 2009, το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού 2010 προβλέπει μικρότερα κονδύλια για την εσωτερική αγορά και την πολιτική, και την πολιτική προστασία των καταναλωτών Παρόλα αυτά, το σχέδιο γενικού προπολογισμού δεν προβλέπει τον ξεχωριστό προπολογισμό που αφορά το Solvit, τη γραμμή προπολογισμού για το Solvit. Ε, για το 2010 έχουν μειωθεί τα κονδύλια ειδικότερα για ε, γραμμές που αφορούν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ε, η γνωμοδότηση ζητεί μία ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού για το Solvit και αύξηση κατά 1 εκατομμύριο ευρώ. Το εκατομμύριο για το εκατομμύριο δεν υπάρχει παρεξήγηση όπως με το δισεκατομμύριο και το τρισεκατομμύριο. Και για τα πιλωτικά προγράμματα που αφορούν ε, την πολιτική καταναλωτών. Αύξηση των σχετικών, σχετικού ποσού σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας πω Καταρχάς ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης λειτουργίας της εσωτερική αγοράς μέσω καλύτερης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τον τομέα των υπηρεσιών και την εφαρμογή της, ε, του κεκτημένου σχετικά με την οδηγία περί υπηρεσιών. Ε, ζητώ επίσης τη συνέχιση ξεχωριστής γραμμής ε, προπολογισμού για το Solvit, όπως επίσης και για την ενίσχυση της αγοράς, εναρμόνιση των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν πληροφορίε και βοηθούν στη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ε, ε, ε, τελωνίων, ε, αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση των ελέγχων στην εξωτερική, στα εξωτερικά σύνορα για την καταπολέμηση της απάτης ε, και του λαθρεμπορίου, αύξηση λοιπόν της αποτελεσματικότητας των τελωνιακών υπηρεσιών. Επίσης υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόθεσή της να εδρεώσει τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει μέσω ενός πίνακα συγκριτικής αξιολόγησης με σκοπό βέβαια ε, την ενίσχυση του μηχανισμού ε, της αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Επίσης, ε, ιδιαίτερη σημασία δίνει στην αύξηση της γνώσης της ε, ε, επιχειρηματικότητας και των οικονομικών. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, στόχο τον οποίο θέλουμε να προωθήσουμε. Επίσης, ε, αποκατάσταση των αρχικών ποσών του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού. Υπήρξαν κάποιες τροπολογίες ε, για την ε, έκθεσή μου, τις οποίες εν μέρη ε, υποστηρίζω και έχω και κάποιες τροπολογίες για την... σε σχέση με αυτά που είχα πει στο, στην ανταλλαγή απόψεων, δηλαδή αύξηση των κονδυλίων για το Solvit και βέβαια ε, βελτίωση των σχετικών ε, ε εγχειρημάτων ε, κατόπιν συζήτησης με τον κύριο Σβάμπ. Επίσης, Ήθελα να σας πω ότι είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και περαιτέρω σχόλια. θα χαρώ να απαντήσω και σε ερωτήσεις. Πρόεδρος. σκιώδεις εισηγητές ε, από τις άλλες ομάδες θέλουν να πάρουν το λόγο. Νομίζω ο κύριος Φάμπη θέλει να πάρει το λόγο, αλλά πρώτα η κυρία Γκέπχαρτ, επειδή απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άλλος σκιώδης ε, εισηγητής ε, ή κάποιος που τον αντικαθιστά για να πάρει το λόγο. Πρώτα η κυρία Γκέπχαρτ. Ο Λουί Γκρέκ ε, είναι ο σκιώδης εισηγητής μας, αλλά εφόσον δεν παρίσταται θα αναλάβω εγώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του ε, και τις προτάσεις που είναι επικοδομητικές και θα ήθελα ιδιαίτερος να τον ευχαριστήσω διότι έχει συμπεριλάβει και ιδέες του τότε σοσιαλιστικού τις τότε σοσιαλιστικές ομάδες οι οποίες τότε είχαν απορριφθεί από το ΕΛΚ και από τους φιλελεύθερους. Βλέπουμε όμως ότι τώρα και οι φιλελεύθεροι και οι χριστιανοδημοκράτες έχουν αποδεχθεί τις προτάσεις μας και μάλιστα έχουν προχωρήσει και πέραν από τις προτάσεις των σοσιαλδημοκρατών και των εκπροσώπων της πολιτικής μου ομάδας. Γι' αυτό και θα υπερψηφίσω με τα μεγάλη χαρά τις προτάσεις σας και ιδίως για τα θέματα τα οποία έχουμε επεξεργαστεί ο Λουί και εγώ διότι ε, βλέπουμε ότι αξίζει να μάχεται κανείς διότι έτσι μπορεί κανείς να πείσει τις άλλες ε, πολιτικές ομάδες ότι το Solvit και το Scoreboard δηλαδή ο πίνακας βαθμολόγησης είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω αρκεί να υπάρχει υπαρκής χρηματοδότηση και γι' αυτό ευχαριστώ ευχαριστώ εν ονόματι τον Λουί, τον οποίο δεν ήθελα να προκαταλάβω, αλλά Λουί πήρα τον λόγο επειδή δεν ήσουν στην αίθουσα, αλλά είσαι, έχεις τη διάθεσή σου αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ευχαριστώ Εύλην. Ο Άντριου Σουάμπ βλέπω ότι μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Η Χάιντι Ρούλε, μήπω θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που ελέγχθησαν, δηλαδή ότι αυξάνεται η γραμμή του προπολογισμού για το Solvit και ευχαρίστω θα την αποδεχθούμε. Ο Άντριος Σφάμπ. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω, τα χαίρομαι που υπάρχει ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτολα και ίσως και κάποιος άλλος προτού παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας ε, για την παρουσίαση των θεμάτων και έχω όμως και μία ερώτηση σχετικά με την στήριξη των οργανώσεων προστασίας του καταναλωτού και ιδίω ε, ε, των ε, νέων κρατών που προσφάτως προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ σημαντική για τη στήριξη της προστασίας των καταναλωτών και μπορέσαμε έτσι να προβάλλουμε το θέμα αυτό. Λόγω όμως της οικονομικής κρίσεως, ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρες, ε, όπου ε, έχει μειωθεί τώρα ο προπολογισμό για την προστασία των ε, καταναλωτών. Θα ήθελα να ξέρω εάν ο εισηγητής μπορεί να μας πει τι έχει γίνει με την μείωση των πιστώσεων και αν πρόκειται να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο όπως πριν από τα πέντε χρόνια. Θα ακούσω τις απόψεις, αλλά θα ήθελα πρώτα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον προπολογισμό, ο David Μέιρ ε, πρόκειται να μιλήσει και δεν ξέρω εάν θεωρεί ότι η γενεοδορία της Επιτροπής αυτής ε, είναι υπέρμετρη, δηλαδή αν θα έχουμε τα χρήματα τα οποία ζητούμε για, εάν συμφωνήσουμε για να προχωρήσουμε. μπορώ να σας πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων που έχετε διατυπώσει ε, διότι πρόκειται για έναν μικρό προπολογισμό ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν και χρειάζεται παρακολούθηση και κατανόηση για να καταλάβουμε πως μια τόσο μεγάλη αγορά για τους καταναλωτές ε, είναι ένα πολύ εκτενές πρόγραμμα. Καλή τύχη λοιπόν. Ωραία. Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας που θέλει να συμπληρώσει ή είσαστε ευτυχοί με την πρόταση. Όχι, ωραία. Λοιπόν, ε, υποθέτω ότι είσαστε όλοι ευτυχείς. Κρίσιαν, θέλεις τότε ε, να μας πεις που βρισκόμαστε σχετικά με την αυριανή ψηφοφορία. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει καλή δουλειά διότι περιμέναμε την πρότασή τους για όλα τα θέματα. Βεβαίως ε, υπάρχει μία χωριστή πρόταση για το Solvit και ε, για την ε, παρακολούθηση των μέτρων. Έρχομαι τώρα στις 12 νέες χώρες ε, διότι είναι πολύ βασικό για την προστασία των καταναλωτών να υπάρχουν προγράμματα όπου μπορούν να υποφεληθούν οι ενώσεις καταναλωτών και γι' αυτό προσπάθησα να διατηρήσω τους ίδιους αριθμούς με πέρυσι παρόλο που εφέτος θα έπρεπε να μιλήσουμε για οικονομική κρίση και ίσως κάποιος θα περιμένει ότι θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα να δαπανηθούν. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της κοινοτικής δράσης και γι' αυτό προσπαθώ να αποκαταστήσω αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όπως είπα στην αρχή, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αύξανε κάπως το ποσό σε σχέση με αυτό το οποίο δαπανήθηκε το 2009. Δεν ξέρω πόσα χρήματα από αυτόν τον προπολογισμό ε, θα ε, αποδοθεί στο πρόγραμμα για τις ε,

Ε, οργανώσεις των ε, καταναλωτών. Διότι ε, για το πρόγραμμα παρακολουθήσεως ζήτησα ορισμένες διευκρινήσεις για τα προγράμματά τους και κάθε χρόνο θέλουν να κάνουν γενικές εκθέσεις για τους καταναλωτές που θα κοστίσουν 1,2 εκατομμύρια και επίσης περαιτέρω μελέτες που θα κοστίσουν 500.000 ευρώ και θα είναι προς όφελος όλων των καταναλωτών και το Solvit που έχει κέντρα σε όλες τις χώρες και διαθέτει διαφορετικές γραμμές πιστώσεων θα μπορέσει να συμβάλλει προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κριστιό εν ονόματι όλων μας που ανέλαβε σε αυτή την εργασία. Οπότε η ψηφοφορία θα είναι αύριο το πρωί και μετά από την παρουσίαση και την συζήτηση με την κυρία Σαβωνή στις 11. Ε, η κυρία Σαβωνή και εγώ θα έχουμε μετά την παρουσίασή της μία συνάντηση με τον τύπο και έτσι ε, θα με αντικαταστήσει μία αντιπρόεδρος και ελπίζουμε ότι όλοι θα είσαστε εδώ αύριο για την ε, πρώτη ψηφοφορία της Επιτροπής αυτής. Κρίσιαν, εσύ ήσουν πολύ δραστήριος ε, εν ονόματί μας γιατί στην προηγούμενη θητεία είχες καταρτήσει ε, διάφορες νομοδοτήσεις για την Επιτροπή Περιβάλλοντος για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία συζητήσαμε σήμερα το πρωί και με τον κύριο Φεχόηγεν σήμερα το απόγευμα μάλλον. Οπότε, ε, μήπως μπορείς να μας ενημερώσεις, διότι έχουμε το κείμενο και θα σου πρότεινα ε, να το παρουσιάσεις και μετά θα ε, παρακαλέσω τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων αν υπάρχουν σχηριώδεις ε, εκπρόσωποι για να μπορέσουν να σχολιάσουν αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, τον Δεκέμβριο 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε ορισμένες προτάσεις οι οποίες είναι γνωστές με την ονομασία φαρμακευτικό πακέτο. Ε, επ' αυτόν πρέπει να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και επειδή έχουμε πολλά νέα μέλη στην Επιτροπή μας, θα ήθελα να επαναλάβω σύντομα ορισμένες παρατηρήσεις που είχα κάνει το Μάρτιο του 2009 στην Επιτροπή αυτή, όταν έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. Έχετε επίσης το έγγραφο εργασίας το οποίο έχω καταρτήσει και αφού ε, καθορίσουμε ε, το χρονοδιάγραμμα θα αναφέρω τα θέματα που θα συζητήσουμε στην Επιτροπή. Αναφερόμαστε εις ε, την ενημέρωση του κοινού για τα φάρμακα όσον αφορά την ιατρική συνταγή και τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα οδηγία. Ξέρετε ότι το θέμα αυτό τώρα ε, ρυθμίζεται από την οδηγία 83 ε, του 2001 ε, όπου αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό 726 του 2004 οι διαδικασίες χορήγησης αδικίες και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα. Θέλουμε λοιπόν τώρα να βελτιώσουμε και να ρυθμίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό για να υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση στη διαδικασία ενημερώσεως των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που προτείνουμε είναι τα εξής. Καταρχήν να διευξηνήσουμε ότι επιτρέπεται ε, να πληροφορούν το κοινό για τα φάρμακα μόνο οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας αυτό όσον αφορά τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή και αναφέρονται σε αυτή την οδηγία. Δεύτερον, να υπάρχουν εναρμονισμένοι όροι όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών που επιτρέπεται να παρέχονται, να θεσπίζονται εναρμονισμένα πρώτα ποιότητα για τι εν λόγω πληροφορίε, να καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι διάβλοι παροχή πληροφοριών. Πέμπτον, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε παρακολούθηση για τι πληροφορίε που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων, ώστε να συνεκτιμάται η διασυνοριακή φύση των πληροφοριών. Χαιρετίζω τις προτάσεις αυτές γιατί πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα εμποδίσουμε τις την παραπληροφόρηση και τις λανθασμένες ε, πληροφορίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτού. Ελπίζω ότι οι θεραπείες ε, θα μπορέσουν επίσης να συμβάλλουν στην βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων ασθενών και ε, ελπίζω ότι θα έχουν καλής ποιότητος ενημέρωση ασχέτως της γλώσσας τους ή της προέλευσής τους. Ε, τώρα υπάρχει μια ιδιάζουσα κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες προσεγγίσεις κατά την εφαρμογή της παλαιάς οδηγίας, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει σε διαφορετικές ρυθμίσεις για διάφορα φάρμακα σε διάφορες αγορές, δηλαδή ε, μια, ένας φαρμακοβιομηχανός δεν μπορεί να δίνει τις ίδιες πληροφορίες σε όλες τις χώρες για τις οποίες έχει άδεια κυκλοφορία των φαρμάκων του και αυτό είναι ιδιάζον διότι θα πρέπει να υπάρχει η ενία ενημέρωση των Ευρωπαίων ασθενών. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες μεταξύ των πολιτών μας. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ εις ε, τις διάβλους παροχής πληροφοριών, διότι υπάρχει μεγάλος ε, σκεπτικισμός για το κατά πόσον η φαρμακοβιομηχανία είναι η σωστή πηγή πληροφοριών, και ε, πολλοί δεν θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για αυτό το λόγο. Εάν όμως υπάρχουν σαφείς κανόνες δεν βλέπω γιατί πρέπει να φοβούμαστε ε, ότι θα υπάρχει ε, κακή χρήση της διαταρότητας αυτός από τη βιομηχανία. Δεν προτείνω βέβαια η βιομηχανία να αποτελέσει την μόνη ε, πηγή μαζί με τις ε, αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει και οι οργανώσεις των ε, καταναλωτών και των ασθενών να συμβάλλουν για να υπάρχει καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Αλλά το πιο βασικό θέμα είναι η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου, διότι ε, βλέπουμε όλο και περισσότερο προσπάθεια ενημερώσεως μέσω του διαδικτύου και θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα μας εγγυώνται ε, την ποιότητα των πληροφοριών που δίνονται μέσω αυτής της οδού. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προκαταρτική εξουσιοδότηση για τις ε, ε, πληροφορίες που δίδονται στο διαδίκτυο ε, αποφεύγοντας ένα γραφειοκρατικό σύστημα και σπατάλη πόρων και, και θα αποφύγουμε και τα προβλήματα για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα από όλες τις απόψεις. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο διαθέσιμο και αναμένω να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων μας. Ευχαριστώ, Κρίστιαν. Πρέπει να σας πω ότι ετοιμάσατε ένα έγγραφο εργασίας ήδη επί του το οποίο ε, είχαμε ήδη δει ε, και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους συναδέλφους αλλά πιστεύουμε ότι σε αυτό θα βασιστείτε για να το βελτιώσετε και θα ήθελα να του στους συναδέλφους ότι Υπάρχουν ε, στις ιστοσελίδες για την ημερήσια διάταξη όλες οι συνδέσεις για να μπορέσετε να ανατρέξετε ε, σε πληροφορίες. Η κυρία Ρόιτοβα είναι ε, σκιώδης εισηγήτρια για το ΕΛΚ και ζητά το λόγο και η κυρία Στήλερ και η κυρία Γκέπχαρτ. Κάποιος άλλος δεν βλέπω, οπότε η κυρία Ρόιτοβα πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Μπουσόη γιατί είναι πολύ εμπαριστατωμένη η προσέγγισή σας του θέματος. Αλλά λείπει μία εξήγηση για κάποιες από τις προτάσεις που σκοπό έχουν την εναρμόνιση. Γιατί στην πράξη, και το έχω δει αυτό, το έχω ελέγξει και εγώ πολλές φορές, Όταν παίρνει κάποιος μία συνταγή από έναν ε, γιατρό σε άλλη χώρα και ας πούμε πάει στο Βέλγιο με τη συνταγή ή πηγαίνει σε, μια, σε ένα φαρμακείο ε, σε μια άλλη χώρα, ο φαρμακοποιός χωρίς κανένα πρόβλημα μπορεί να βρει ποιο είναι το περιεχόμενο του φαρμάκου. γιατί υπάρχει μια σχετική βάση δεδομένων και αν αυτό το φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί ο φαρμακοποιός να προτείνει ένα διαφορετικής ονομασίας φάρμακο, το οποίο όμως έχει τα ίδια ε, συστατικά. Αυτό το σύστημα λειτουργεί και στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες και θα ήθελα να μάθω κατά πόσο υπάρχουν χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις οποίες θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόβλημα Ε, με αυτό το σύστημα. Οι φαρμακοποιοί μου εξηγούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως πρόβλημα με κάποια... με κάποια βοηθήματα. Μήπως θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο για ιατρικά βοηθήματα και λιγότερο για ε, σκευάσματα Οι ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πρόβλημα πρόσβασης στα φάρμακα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι, σε λίγο θα απαντήσει η Επιτροπή στο ερώτημα αυτό. Αλλά πρώτα η κυρία Στήλερ και η κυρία Γκέπχαρτ. Thank you. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόταση του κυρίου Μπούσο και εγώ έχω εργαστεί επί του θέματος αυτό όταν ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και για το φαρμακευτικό πακέτο. Κανένας δεν διαφωνεί ότι όλοι θέλουμε, θέλουμε οι ασθενείς ε, να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη ε, πρόσβαση στις πληροφορίες και μου έκανε εντύπωση όταν είπατε ότι υπάρχει ε, μια τάση ενημέρωσης για τα φάρμακα. Ναι, αλλά η φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να πουλήσει και τα ε, φάρμακά της, οπότε πρέπει να δούμε πώς η ενημέρωση θα είναι η σωστή. Στο παρελθόν έχω εργαστεί όσον αφορά, έχω εργαστεί για, τη, για την συσκευασία των φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν μιλούσε καθόλου για θέματα αναπηριών, για άτομα με αναπηρίες. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουν όλοι πρόσβαση ε, στην ενημέρωση αυτή, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που ενδεχομένω δεν χρησιμοποιούν το ίντερνετ και πρέπει όλοι με ισότιμο τρόπο να μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, στην ενημέρωση αυτή. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ χωρίς διακοπή μπορώ να συνεχίσω τα επιχειρήματα της Κατρίν. Και εγώ θα ήθελα ακριβώς αυτό το πρόβλημα της ποιότητας της πληροφόρησης ε, να εξετάσουμε σε βάθος. Και αυτή η τοποθέτηση με εξέπληξε ότι η φαρμακοβιομηχανία λέει είναι εκείνη που γνωρίζει καλύτερα ποια πληροφόρηση μπορεί να δοθεί και τι πρέπει να λέει. Το βρίσκω πολύ προβληματικό αυτό. Φυσικά γνωρίζει καλύτερα τα προϊόντα της η φαρμακοβιομηχανία, όμως έχει και το μεγαλύτερο συμφέρον να πωλήσει, να, να πουλάει αυτά τα φαρμακευτικά της προϊόντα. Και γι' αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε σε βάθος και να δούμε μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε επίσης ότι όλα τα φάρμακα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά πρέπει σίγουρα πάντα να εξετάζονται πιο πριν και να διοδοτούνται από κλινικές, από τμήματα έρευνας πανεπιστημίων και ίσως πρέπει και αυτοί να εμπλέκονται για τα θέματα πληροφόρησης που πρέπει να δίνονται πληροφόρηση που πρέπει να δίνετε. Η ποιότητα είναι σημαντικό θέμα, πρέπει να μας ξαναπροβληματίσει, να δούμε τι θα κάνουμε για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο και άλλο είναι όσον αφορά την ποιότητα των διαχειωμένων πληροφοριών. Πέρα από αυτό, ο τρόπος με τον οποίο συντάσσονται οι πληροφορίες αυτές, ώστε να είναι εύληπτες και κατανοητές για τους πολίτες. Εχθές διάβασα κάτι. Και όχι σε σχέση με αυτήν την έκθεση εδώ, αλλά το κείμενο το διάβασα τρεις φορές για να το καταλάβω. Ήταν στα γερμανικά και δεν το καταλάβαινα. Τρεις φορές έπρεπε να το ξαναδιαβάσω, διότι ήταν τόσο γεμάτο ε, ειδική ορολογία που δεν μπορούσα να το, να το κατανοήσω ε, εύκολα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα της, ε, του εύληπτου κατανοητού χαρακτήρα από τους πολίτες και να το ρυθμίσουμε σχετικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που ανέφερε πιο πριν η Κατρίν, η, η συνάδελφος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ασθενείς στην Ευρώπη χρειάζονται καλύτερες πληροφορίες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν καλύτερες πληροφορίες για τα φάρμακα που τους δίνονται ή θα έπρεπε να τους δίνουν. Το πρόβλημα είναι ποιος θα τους δώσει αυτές τις πληροφορίες στους πολίτες. Για μένα έχει, έχει τεράστια σημασία να είναι ανεξάρτητος ο φορέας, ο θεσμός που θα πληροφορεί τους πολίτες. Δηλαδή κάποιος που δεν θα αποκομίζει κέρδος από το ότι σε ασθενείς θα χορηγούνται φάρμακα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι την πρόταση θα πρέπει να την εξετάσουμε να δούμε αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, αυθεντική ανάγκη κάτι να αλλάξει σε σχέση με σημερινή πρακτική και να διαρωτηθούμε πώς θα μπορέσουν οι γιατροί να εμπλέκονται που συνταγογραφούν κάποια, πράγματα, κάποια φάρμακα και να εμπλέκονται περισσότερο. Θα πρέπει περισσότερο να εξετάσουμε σε βάθος αυτή την πρόταση. Δεν νομίζω ότι βρήκαμε σωστή ισορροπία ακόμα. Uh, Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη μου παρέμβαση επιτρέψτε μου να συγχαρώ και να συγχαρώ τον πρόεδρο και τους συναδέφους με αυτήν την πρώτη μου παρέμβαση που ξεκινώ έτσι. Η λειτουργεί η διερμηνία, είναι όλα εντάξει, ωραία εντάξει λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπουσόη για τη δουλειά που έχει κάνει. Είναι χωρίς αμφιβολία πολύ σοβαρή αυτή η δουλειά, αυτό το σημείο. Και όπως υπογραμμίστηκε από τις διαφορετικές παρεμβάσεις πιο πριν, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο να ρυθμιστεί σωστά. Φυσικά είναι επίσης ένα κατεπήγον θέμα, έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα. Γιατί, Γιατί όλοι μας είμαστε καταναλωτές και μας κατακλίζει, μας πλημμυρίζουν με πληροφορίες που δεν είναι πάντα οι πιο τέλειες και δεν υπάρχει σωστή ισορροπία και πολλές φορές είναι αμφισβητήσιμες αυτές τις πληροφορίες. Πολλές φορές ε, υπάρχει περιττή πληροφόρηση, το spam που μας περνάει μέσω από τους υπολογιστές μας, ε, περιττές ε, διαφημίσεις, πληροφορίες και δεν ξέρουμε τι πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ, μεταξύ του στάριου και της ήρας. Όμως εδώ είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών, να αναβαθμιστεί. Είναι φυσικό, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στις χώρες μας, πολλές διαφορετικές μέθοδοι ενημέρωσης των πολιτών. Υπάρχει παραδοσιακή συμβατική μέθοδος, ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει μέσα στο πακέτο, στη συσκευασία του σκευάσματος. Στην Πορτογαλία είναι μπούλαρτο αυτό το, ε, ε, η πληροφόρηση, οι οδηγίες χρήσης φαρμάκου και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να διαβαστεί αυτό το κείμενο και να γίνει κατανοητό από τους πολίτες. Λοιπόν, δεν πρόκειται εδώ απλά και μόνο για μια, α, ας το πω έτσι, εξαπλούστευση ενός περίπλοκου θέματος. Ίσως θα είναι αδύνατο κάτι τέτοιο και πολύ δύσκολο. Αυτό όμως που θέλουμε να πετύχουμε εδώ και ζητούμε είναι να βρούμε ένα μηχανισμό, μηχανισμούς, ώστε ανεξάρτητη πληροφόρηση να είναι διαθέσιμη στους πολίτες και προσβάσιμη, προσπελάσιμη στους καταναλωτές. Και εδώ έχουμε πρόβλημα ακριβώς. Εδώ εδώ έχουμε ένα πρόβλημα για το, τη διαφοροποίηση μεταξύ της έννοιας πληροφόρησης και της έννοιας της διαφήμισης, η προαγωγής ε, προϊόντος. Αν δεν είναι ανεξάρτητη η πληροφόρηση, γίνεται προαγωγή, διαφήμιση προϊόντος. Εντάξει, ο μηχανισμός, ο μοναδικός μηχανισμός για να έχουμε πληροφόρηση ανεξάρτητη είναι να βρούμε μια συνένεση, να πετύχουμε μια συνένεση μεταξύ τριών εταίρων. Φυσικά οι ρυθμιστές, το κράτος που πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος ε, της, ε, του λογαριασμού των φαρμακευτικών δαπανών, 60, 70 ή 80% των δαπανών για την φαρμακευτική κάλυψη στις χώρες μας, φυσικά από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής που χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να ξέρει τι του γίνεται παρότι η ανάγκη του φυσικά είναι, χειρίζεται μέσω, ε, αντιμετωπίζεται μέσω του ιατρού, μέσω της σχέσης που έχει με τον γιατρό του ο ασθενής και φυσικά έχουμε και τη βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία που ε, ακολουθεί την καινοτομία όλο και περισσότερο καινοτομή και παράγει προϊόντα. Αυτό θέλω να πω ότι είναι απαραίτητη αυτή η δουλειά και πρέπει να την κάνουμε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Πρέπει όμως να βρούμε ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει να διαχέεται ανεξάρτητη πληροφορία. Και επιμένω εμένω σε αυτό. Για αυτή την ανεξάρτητη πληροφόρηση πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Θα είναι το βρετανικό πρότυπο που φαίνεται να λειτουργεί καλά. Θα είναι το σουηδικό πρότυπο που και αυτό φαίνεται να έχει καλά επιχειρήματα υπέρ αυτού. Δεν το ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι. Αλλά αυτό το θέμα πρέπει να τύχει πολλή προσοχή. Να εμβαθύνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. I, I meant Ευχαριστώ. Ήθελα επίση να σα καλωσορίσω και στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την, διορατική ορατική σα αυτή παρέμβαση. Θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο πριν uh, ο κύριο Στίβεργκερ από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων uh, λάβει το λόγο, γιατί τον ενδιαφέρει ιδιαίτερο αυτή η πρόταση, να απαντήσει ενδεχομένω και σε κάποια σχόλια. Και μετά θα δώσω το λόγο και στον κύριο Μπουσόη να ε, συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση και τη γενική υποστήριξη στην πρόταση της Επιτροπής. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε την πρόταση αυτή, αφού τη βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Κατόπιν όσων άκουσα, θα ήθελα να απαντήσω καταρχάς όσον αφορά την ισορροπία της, ε, στη βιομηχανία ότι έχει δηλαδή συμφέρον να ε, πουλήσει περισσότερα προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να ε, μας απασχολήσει. Δηλαδή αφορά κυρίως ε, η νομοθεσία αυτή την κάλυψη ενός νομικού κενού. Το λέω αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεύτερον, θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ενημέρωσης. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής. Ε, να υπάρχουν κριτήρια ποιότητας τα οποία ε, πρέπει να πληρεί η φαρμακευτική ε, βιομηχανία. Δεν θέλουμε να υπάρχει μονοπόλιο του κλάδου, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες από όλους τους εταίρους ε, συμπεριλαμβανομένων των ε, αρμοδίων αρχών για να συμπεριλάβουμε το απαραίτητο επίπεδο πληροφοριών ε, για τους ασθενείς. Στην ε, εν λόγω πρόταση επικεντρωνόμαστε κυρίως σε αυτά τα οποία επιτρέπει ο κλάδος και ε, σε αυτά τα οποία δεν πρέπει να επιτρέπονται και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο την ομοθεσία περί ε, φαρμακευτικών. Θέλουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές και έχουμε στο φαρμακευτικό πακέτο περισσότερες πληροφορίες από αυτού. Τώρα όσον αφορά το θέμα των αναπηριών θα ήθελα να για το άρθρο 110 ε, F ε, που μιλά ε, ειδικότερα για την ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν τα φάρμακα. Είναι ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα. Επίσης η πρόσβαση των ασθενειών, των φαρμάκων, η πρόσβαση στα φάρμακα ορισμένων ασθενών σε ορισμένες χώρες. Αναφέρθηκε αυτό το θέμα του υποκατάστατου φαρμάκου, δηλαδή αν μπορεί να υποκαταστήσει ο φαρμακοποιός ε, ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει με ένα άλλο φάρμακο το οποίο έχει στη διάθεσή του. Σε μερικές χώρες είναι, ε, έχουν αδειοδοτηθεί κάποια φάρμακα και σε κάποιες χώρες όχι, αλλά για παράδειγμα, μπορεί σε μία χώρα να έχει διατεθεί ε, το ε, φάρμακο από την φαρμακευτική ε, εταιρεία και στην άλλη όχι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα ε, πρόσβασης και αυτό το έχουμε, το έχουμε συμπεριλάβει σε κάποιες από τις ανακοινώσεις μας, ε, κάτι το οποίο αφορά και το μέλλον ε, του φαρμακευτικού πακέτου και το μέλλον της φαρμακοβιομηχανίας βεβαίως. Υπάρχουν κάποια προβλήματα λοιπόν πρόσβασης σε κάποια φάρμακα σε κάποιες χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, uh, Και εγώ ε, σας ευχαριστώ για αυτήν την πάρα πολύ σαφή ε, εξήγηση του ιστορικού. Κριστιαν, θέλεις να συνοψίσεις και να μας δώσεις ε, και κάποια ένδειξη του χρονοδιαγράμματος. Καταλαβαίνω βέβαια ότι περιμένεις και την περιτροβή περιβάλλοντος, αλλά μήπως μπορείς να μας πεις περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, Μάλκολ. Θα ήθελα να πω μερικά ε, πράγματα και εγώ, θα είμαι σύντομος. Η πρόταση της Επιτροπής ε, και βέβαια και από αυτά που είπα. Δεν είπα ότι η φαρμακευτική βιομηχανία θα είναι η μόνη πηγή πληροφοριών. Απλώς πιστεύω πραγματικά ότι δεν πρέπει να εξαιρέσουμε την πηγή αυτή. Μιλάμε βέβαια και για τις εθνικές αρμόδιες αρχές ε, οι οποίες θα παραμείνουν υπεύθυνε για τον έλεγχο, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγουν ε, οι ε, ενώσεις ασθενών, ιατρική σύλλογη. Είτε μιλάμε λοιπόν, πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα, τον οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε όπως προτάθηκε, είτε πρόκειται για τη φαρμακευτική βιομηχανία, νομίζουμε ότι οι πηγέ είναι σημαντικέ και μπορεί να μα βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματα. Η κατάσταση λοιπόν είναι διαφορετική. Ε, υπάρχει ένα μοντέλο στις βόρειες χώρες, ένα άλλο μοντέλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσης μου αρέσει πολύ, ένα διαφορετικό μοντέλο στην Πορτογαλία, ένα διαφορετικό μοντέλο στα νέα κράτη-μέλη. Οπότε η βασική πρόθεσή μας είναι να εναρμονίσουμε όλα αυτά τα μοντέλα και να, υπάρχει, ε, υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές σε σχέση με την πληροφόρηση ε, των ασθενών και την πρόσβασή του στις πληροφορίες αυτές και νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να το οργανώσουμε αυτό. Τώρα όσον αφορά τη διαφήμιση για τα, ε, για τα φάρμακα ε, που χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης πρέπει να παραμείνει η απαγόρευση. Δεν ξέρουμε ειδικότερα πού είναι η διαφήμιση και πού είναι η ενημέρωση και εγώ δεν θέλω να ενισχύσω κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να προωθηθεί αυτή η ιδέα επουδενή. Αλλά το να βρούμε το όριο δεν είναι εύκολο. Ε, και πάντοτε είναι ένα πολύ ευαίσθητο ε, θέμα και διαφιλονικούμενο. Ποιο είναι το διαχωριστικό όριο μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση παρόλα αυτά. Κάτι ακόμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα για να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ να προτείνω χρονοδιάγραμμα γιατί πρέπει να περιμένουμε την πρόταση του, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δεν θέλω λοιπόν να προτρέξω, ε, ούτε θέλω να βιαστούμε. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε με ε, λεπτομέρειες αυτό το πολύ, αυτή την πολύ σημαντική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ε, γιατί ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Έχουμε και ένα έγγραφο όσο από το Μάρτιο και θα το ε, διανύμουμε εκ, μέρου, νέου. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής για τα σχόλιά τους. Η ε, δεξίωση της Σουηδικής Προεδρίας μας περιμένει και τα ποτά μας. Έχουμε επίση και το θέμα το οποίο είχε αναλάβει ο κύριος Αγγελάκα, ο οποίο δεν επανεξελέγει και αφορά επίση το φαρμακευτικό πακέτο, δηλαδή τα παραποιημένα ε, ιατρικά προϊόντα. Δεν έχουμε πληροφορίες, ε, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να το παρουσιάσει τώρα. Προτείνω να έχουμε μία συζήτηση σε κάποια μελλοντική ημερομηνία όταν θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ε, ότι θα αποφασίσουν οι συντονιστές ποιος θα αναλάβει την έκθεση αυτή και πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε περαιτέρω. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και κυρίως τα νέα μέλη της Επιτροπής μας ε, που ε, συνέβαλαν στη συζήτηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θέλετε τόσο πολύ να συμμετέχετε στις συζητήσεις μας και το δείξετε. Θα ξανασυναντηθούμε αύριο το πρωί 9 η ώρα για το πρώτο τμήμα των συζητήσεών μας ε, για, τα, ε, για την ε, ετικετοθεσία των προϊόντων κλωστοφαντουργίας και θα έχουμε και μία συζήτηση για τον προϋπολογισμό και μετά μία ενημέρωση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα υπάρξει λοιπόν, θα γίνει μια συζήτηση κατατοπιστική για να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Γεια σας.